χρειάζεται να επανερχόμεθα σε θέματα αυτά και αντίθετα να εστιάσουμε την προσοχή μας στην έρευνα και την καινοτομία. Σας ευχαριστώ, λέει και ο Πρόεδρος, κυρία Πρόεδρε του Συμβουλίου και τον κύριο Αντιπρόεδρο, κύριο Σεφκοβιτς. Κλείνει η συζήτηση λοιπόν για το θέμα αυτό. Περνάμε στο επόμενο σημείο της συζήτησής μας σήμερα είναι η δήλωση της Αντιπροέδρου της Κομισιόν και υπά του της εκπροσώπου για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας σε σχέση με την κατάσταση στη Μεσόγειο, ιδίως στην την, Ισία και στην Αίγυπτο. Κυρία Αντιπρόεδρε και υπάτη εκπρόσωπε, καλωσορίσατε στο κοινοβούλιο μας. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτέ, μετά τα πρόσφατα γεγονότα στην Τινησία και μετά και στην Αίγυπτο, είδα ότι οι λαοί και των δύο χωρών είχαν πολλούς λόγους απελπισίας αλλά και λόγους να ελπίζουν στους εταίρους τους. Το μήνυμα είναι σαφές. Τα πολιτικά του συστήματα δεν μπορούσαν πια να λειτουργήσουν και πρέπει να συμβεί αλλαγή. Εκφράζω την, ε, το θαυμασμό μου για το θάρρος τους. Ιδιαίτερα καλό για πνεύμα ηρεμίας και συμφιλίωσης. Θα μιλήσω πρώτα για την Τινησία. Οι αλλαγές εκεί είναι αξιοσημείωτες και άνοιξαν το δρόμο για περισσότερο εκδημοκρατισμό της χώρας, για εκδημοκρατισμό μάλλον της χώρας. Έχουν γίνει προσπάθειες για να αντιμετωπιστούν τα αιτήματα του λαού. Η μεταβατική κυβέρνηση έχει λάβει ορισμένα μέτρα όπως απελευθέρωση πολιτικών κρατουμένων, διασφάλιση της ελεύθερης έκφρασης και ζήτησε δίκη για τον πρώην πρόεδρο. Έχουν δημιουργηθεί ανεξάρτητες επιτροπές για να τα επιτύχουν όλα αυτά. Η Επιτροπή για την Έρευνα κατά της Διαφθοράς και Δωροδοκίας θα ερευνήσει τα πράγματα και τα τελευταία γεγονότα και σημείωσα επίσης ότι η κυβέρνηση έχει την υποστήριξη των κυρίων αντιπολιτευτικών κομμάτων και συνδικάτων. Η ειρήνευση και η σταθερότητα είναι σημαντική για να μπορέσει την Ισία να κινηθεί προς τη διοργάνωση ελεύθερων και διαφανών εκλογών η Ευρωπαϊκή Ένωση θα στηρίξει τη χώρα και το λαό της σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Και έχουμε ήδη ανταποκριθεί αμέσως. Όχι για να επιβάλλουμε τις δικές μας ιδέες, αλλά για να προσφέρουμε τη βοήθειά μας και τη συνεργασία μας. Την περασμένη εβδομάδα μίλησα με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιουνές, μετά το διορισμό του και συναντηθήκαμε και σήμερα στις Βρυξέλλες. Είχαμε ουσιαστική συζήτηση εδώ που είναι η πρώτη του επίσκεψη εκτός της νησίας από την αλλαγή. Μου επιβεβαίωσε ότι ζητιέται βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά την προπαρασκευαστική φάση τον εκλογών και είμαστε έτοιμοι να στείλουμε μία αποστολή εμπειρογνωμόνων για να δώσει νομικές συμβουλές στις μεταβατικές αρχές για τη διοργάνωση των εκλογών. Την περασμένη εβδομάδα επίσης στείλαμε εκπρόσωπο να συζητήσει εκεί τις ανάγκες του λαού. Αυξάνουμε ήδη το ποσό που χορηγούμε ως βοήθεια και ως και διοργανώνουμε ένα πρόγραμμα πρόσθετης βοήθειας για άμεση ανακούφιση του λαού. Θα αναθεωρήσουμε λοιπόν μαζί με την Τινησία τις προτεραιότητές μας για να λάβουμε υπόψη μας όπως πρέπει τη νέα κατάσταση και να προσαρμόσουμε τα προγράμματά μας. Ο Υπουργός μου ανέφερε σήμερα και ορισμένα σχέδια που έχουν στην Τινησία για διάλογο στις εξής, στους εξής τομείς εκλογική βοήθεια, πέρασμα προς τη δημοκρατία, στήριξη των μη κυβερνητικών οργανώσεων και της κοινωνίας των πολιτών, ένομη τάξη πολέμηση της διαφθοράς και στήριξη των ασθενέστερων οικονομικά περιφερειών της Τινησίας. Επίσης, μαζί με όλα τα κράτη-μέλη, θα δούμε το θέμα περισσότερης και ευκολότερης πρόσβασης στην αγορά μας της Τινησίας. Ο διάλογος θα συνεχιστεί. Θα πάω και εγώ στην Τινησία τη μεθεπόμενη εβδομάδα. Όσο για τα αιτήματα των αρχών της Τινησίας να παγώσουν οι λογαριασμοί του Μπεναλή, αυτά τα βήματα έχουν ήδη αναλυφθεί και τη Δευτέρα το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών θα συζητήσει ακριβώς αυτό το θέμα του παγώματος της περιουσίας των λογαριασμών παραγόντων της παλαιάς κατάστασης. κατάστασης. Σας είχα πει και την περασμένη εβδομάδα ότι στείλαμε έναν διευθυντή στην Τινησία για να συζητήσει με τους προέδρους των επιτροπών που έχουν συσταθεί εκεί τι λύσεις μπορεί να είναι οι καλύτερες. Θα ήθελα να καλωσορίσω εδώ την ε, πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να στείλει και εκείνο αντιπροσωπεία στην Τινησία γιατί είναι κάτι που χρειάζεται. σε αυτήν την ε, δύσκολη στιγμή της μετάβασης προς τη δημοκρατία. Πρέπει να ενδυναμώσουμε όλους τους παράγοντες και τα στοιχεία της κοινωνίας των πολιτών και μη κυβερνητικέ οργανώσεις καθώς και να ενδυναμώσουμε τις φοιτητικέ ανταλλαγέ, Έχουμε τώρα δυνατότητα για αυξημένες εταιρικέ σχέσεις με την Τινησία. Ελπίζω να μπορέσουμε να οικοδομήσουμε αμοιβαίο σεβασμό και περισσότερη συνεργασία, σταθερότητα και δημοκρατικό μέλλον. Και γι' αυτό προσδοκώ ιδιαίτερα στη διοργάνωση των ελεύθερων εκλογών εκεί και την νέα κυβέρνηση. Όταν θα υπάρξει η νέα κυβέρνηση θα έχουμε φυσικά και νέες διαπραγματεύσεις και τέλος ο υπουργό σήμερα μου είπε ότι στην Τινησία έχουν αρχίσει ήδη οι κινήσεις συμφιλίωσης. Ελπίζω να συμφωνείτε ότι αξίζει η Τινησία να κινηθεί προς την κατεύθυνση αυτή. Και τώρα θα μιλήσω για την Αίγυπτο. Πριν από μια εβδομάδα μόλις είδαμε εκεί να σημειώνονται οι πρώτες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που είχαν εμπνευστεί βέβαια από την Δυνήσια και μέσω των κοινωνικών ε, ηλεκτρονικών μέσων έγιναν οι συνεννοήσεις και κατέληξαν σε ολόκληρη εξέγερση σε όλη την Αίγυπτο. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι όλων των ηλικιών και φίλων βγήκαν στους δρόμους και ζήτησαν, απίτησαν τα κοινωνικά τους και οικονομικά τους δικαιώματα στο Σουέ, στην Αλεξάνδρεια, στο Κάιρο και αλλού. Και όλο και διογκωνόταν οι διαδηλώσεις ζητώντας αλλαγή του καθεστώτος και σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας. Οι ειρηνικές με αυτές διαδηλώσεις δέχτηκαν και κάποιες βίαιες επιθέσεις. Χρησιμοποιήθηκε σε πολλές περιπτώσεις, χρησιμοποιήθηκαν σφαίρες από την αστυνομία και το στρατό. Σκεφτόμαστε ιδιαίτερα εκείνους που έχασαν αγαπημένα τους πρόσωπα. Επίσης συνέβησαν πολλές συλλήψεις και ζητούμε από όλα τα κόμματα να αυτοσυγκράτηση. Ζητούμε λοιπόν από τις Αιγυπτιακές αρχές να απελευθερώσουν αμέσως όλους τους κρατούμενους απλούς διαδηλωτές και διαδηλώτριες. Η ελευθερία της έκφρασης είναι θεμελιώδες δικαίωμα του καθενός και της καθεμιάς. Η επιβολή περιορισμών στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στο ίντερνετ είναι κάτι απαράδεκτο και ζητούμε από τις Αιγυπτιακές Αρχές να τις καταργήσουν. Από τις πανεθνικές αυτές διαδηλώσεις ο Αιγυπτιακός λαός έδειξε ότι ζητάει αλλαγή. Εκατοντάδες χιλιάδων σε κάθε διαδήλωση και είναι πάρα πολύ σημαντικό οι φωνές αυτές να ακουστούν. Χρειάζονται τώρα βέβαια συγκεκριμένα μέτρα ήρθε πια ο καιρός για την μετάβαση στη δημοκρατία. Οι αρχές πρέπει να πάρουν στα σοβαρά το θέμα ενός πραγματικού διαλόγου με τις αντιπολιτευτικές αυτές φωνές. Οι Αιγυπτιακές αρχές πρέπει να βιαστούν αν θέλουν πράγματι να υπάρξει μία αληθινή δημοκρατική μετάβαση και να διοργανωθούν ελεύθερες εκλογές. Εμείς προσφέρουμε την πλήρη μας υποστήριξη στην αλλαγή αυτή ώστε να γίνει η Αίγυπτος πιο πλουραλιστική και πιο δημοκρατική. Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι να ενδυναμωθούν τα μέσα που ήδη διαθέτουμε και χορηγούμε για οικονομικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις συνεργασία στον τομέα της ένωμης τάξης, της δημοκρατία του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κυρίες και κύριοι, για μένα η πολιτική είναι θέμα αλλαγής των πραγμάτων και δυνατότητας του λαού να πάρει την τύχη του στα χέρια του με βάση τα αιτήματά του. Δίνουμε λοιπόν, προσφέρουμε στο λαό της Αιγύπτου την πλήρη μας υποστήριξη και αλληλεγγύη γιατί εμείς είμαστε Ένωση Δημοκρατιών. Στηρίζουμε λοιπόν την αλλαγή και συγχαίρουμε το θάρρος του λαού. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Ήπετη εκπρόσωπο. Εκ μέρους της ομάδας του Λαϊκού Κόμματος, ο κύριος Σαλαφράνκα για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Αντιπρόεδρε, ανεξαρτήτως των εξελίξεων και ανεξαρτήτως κυρίως της κατάληξης αυτών των εξελίξεων μπορούμε ήδη να μιλάμε για ένα πριν τα γεγονότα ενώ και ένα μετά τα γεγονότα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της νέες και ταυτόχρονα αυτό θα πρέπει να το κάνει με μία φωνή θα πρέπει να αποφύγει την λεγόμενη κακοφωνία και γι' αυτό ακριβώς δημιουργήθηκε για τέτοιες περιπτώσεις η υπηρεσία σας. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσετε να μας βγάλετε από αυτήν την πολιτική ανοχής θα έλεγα την οποία δείχνουμε απέναντι σε ορισμένους γείτονες ξεκινώντας από τη Λευκορωσία και περνώντας στην νότια πλευρά της Μεσογείου. Απαιτείται περισσότερη δημοκρατία, απαιτείται περισσότερη ε, ελευθερία. Το θέμα είναι λοιπόν μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα τι θα κάνουμε και κυρίως τι θα κάνουμε τώρα. Κυρία Άστον, πράγματι σωστά είπατε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να στηρίξει τις διαδικασίες μετάβασης είναι συμφέρον μας αλλά και υποχρέωσή μας να προειδοποιήσουμε για τους κινδύνους βέβαια που μπορεί να δημιουργήσουν οι διαδικασίες αυτές. Δεν θα πρέπει οι τελευταίες αυτές εξελίξεις να πέσουν όμοιροι θα έλεγα κάποιων διαφορετικών πολιτικών απόψεων. Όπως έλεγε και ο Επίτροπος Φίλεχτες, θα πρέπει να αποφύγουμε τις διαφοροποιήσεις απέναντι στα προβλήματα, στη συγκεκριμένη περίπτωση και ταυτόχρονα θα πρέπει να απαλλαγούμε από τους δημίους που ταλαιπώρησαν τους λαούς αυτούς. Uh, Κύριε Πρόεδρε, κυρία είπατε εκπρόσωπε, συνάδελφοι, τα πρόσφατα γεγονότα στην Τινεσία, στην Αίγυπτο, στην Ιορδανία και αλλού στην περιοχή μας θυμίζουν ότι η ελευθερία δεν είναι απλό, η της ελευθερίας είναι μια βίωτη πραγματικότητα. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι μια κοινωνική επανάσταση, η ε, αναταραχή είναι μια εγγύηση για την αλλαγή αλλά όχι σίγουρα προς το καλύτερο και ελπίζω ότι θα βρούμε μια έμπνευση ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε σε αυτή τη διαδικασία ώστε να είναι μια αλλαγή προς το καλύτερο και όχι πιο στο χειρότερο. Η ανάλυση στην και, για την Τινησία και την Αίγυπτο χρειάζονται, γιατί πρέπει να καταλάβουμε αν κάναμε τα κατά, σωστά πράγματα στο παρελθόν ώστε να αποφευθούν οι κρίσεις αυτές. Ποια είναι τα βήματα που θα πρέπει να κάνουμε στο μέλλον ώστε να προβλέψουμε ή να αποφύγουμε παρόμοιες κρίσεις. Και τέλος, τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να εξασφαλίσουμε ότι οι σημερινές κρίσεις θα οδηγήσουν ε, τα πράγματα προς την ελευθερία για τους εν λόγω λαούς και τη σταθερότητα στην περιοχή. και θα αποφευθεί η περισσότερη αστάθεια ή άλλο είδος αστάθειας ή άλλο είδος ε, απολυταρχισμού ή καταπίεσης. Πρέπει να υιοθετήσουμε μια προληπτική και δραστήρια στάση ως προς αυτό και αυτό σημαίνει στρατηγική. Σίγουρα τα μηνύματά μας ήταν σωστά όταν ε, μιλούσαμε για μεταρρύθμιση και τάξη σταθερότητα. Αλλά ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες και όντως πολλοί από εμά φοβόμαστε γιατί δεν εξετάσαμε αυτέ τι λεπτομέρειε και δεν δείξαμε αρκετή οραματικότητα και ισχύ στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων. Αυτό θα πρέπει να φανεί και στην ικανότητά μα να συνομιλήσουμε με όλου του ε, πλεκόμενου φορεί συμπεριλαμβανομένων των Ισλαμικών δυνάμεων ώστε να μπορέσουμε να του εντάξουμε όλου σε μια θετική διαδικασία. Ελπίζουμε πω η Κομισιόν και το Συμβούλιο θα μπορέσουν να σχηματίσουν μια τέτοια στρατηγική για το μέλλον και θα θέλαμε να ακούσουμε περισσότερα γι' αυτό από εσά. Euh, Μάλιστα κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι αυτά τα οποία ζούμε αυτή τη στιγμή κυρίως στην Τινησία και στις τελευταίες ώρες στην Αίγυπτο είναι ιστορική σημασία αλλά ταυτόχρονα και πολύ τραγικά. Όταν ακούμε τώρα πως υπάρχουν εκατοντάδες εκατοντάδων τραυματίες ε, τις, τις τελευταίες μόλις ώρες και αυτό με κάνει να το σκέφτομαι γιατί βλέπω μια ομοιότητα ανάμεσα στα όσα συμβαίνουν τώρα στη Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Ευρώπη με τα όσα συνέβησαν στην Ευρώπη το 1989 και ακριβώς για αυτό το λόγο θα πρέπει να σας πω εγώ είμαι έκπληκτος αλλά και απογοητευμένος για τον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη κάνει και πάλι τα ίδια ακριβώς σφάλματα που έκανε το 1989. Είναι απίστευτο. Κύριε Πρόεδρε, εμείς η υποτιθέμενη δημοκρατική Ήπειρος δεν έχουμε ακόμα καταφέρει να στηρίξουμε ανεπιφύλακτα τις μάζες, τους λαούς που έχουν κατέβει στον δρόμο και που δεν ζητούν τίποτα άλλο από την υποστήριξή μας. Την στήριξή μας. Και αυτό αγαπητοί συνάδελφοι δεν τα άκουσα ούτε χθες ούτε σήμερα. Ούτε χθες ούτε σήμερα. Από την είπατε εκπρόσωπο. Γιατί κυρία στον Ευρώπη αντιδρά με τόσο αδύναμο τρόπο. Δηλαδή στην πράξη δεν αντιδράσαμε καν. Εσείς αντιδράσατε μετά η Γερμανία, η Γαλλία, η Αγγλία, ε, ξέδωσαν κάποια ανακοινοθέντα ασενάρτητα. Λες και η Ευρώπη δεν υπήρχε. Δεν υπάρχει και πρέπει να σας πω ότι η μόνη σωστή παρέμβαση ευρωπαϊκή ήρθε εκτός Ένωσης. Δηλαδή από τον Τούρκο Πρωθυπουργό, τον κύριο Ερντογάν, που είπε στον Μουμπάρακ ότι πρέπει να ακούσει τις απαιτήσει του λαού του και ότι άρα πρέπει να φύγει. Ήταν η μόνη σωστή αντίδραση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πιστεύω λοιπόν ότι η ανακοίνωση που κάνετε τώρα είναι πολύ σημαντική για αυτούς που είναι στο δρόμο και που αγωνίζονται με τίμημα ίσως και την ίδια τους τη ζωή. Εγώ πιστεύω πως δύο σφάλματα έχουν γίνει από την Ευρώπη τα τελευταίε μέρες. Καταρχήν δεν, καταλα... δεν φαίνεται να έχει γίνει κατανοητό ότι ζούμε ιστορικές ε, στιγμές και ακόμα πιο σημαντικό είναι ότι γίνεται λάθος ανάλυση της κατάστασης. Φοβούμαστε και γι' αυτό υπάρχουν αυτά τα λανθασμένα ανακοινοθέντα. Φοβόμαστε μήπω εγκατασταθεί Ισλαμικό καθεστώ μετά από τι εκλογέ. Εγώ σα το λέω, δεν φοβάμαι. Εγώ εμπιστεύομαι τον λαό τη Τινησία και τον λαό τη Αιγύπτου επιθυμούν τη δημοκρατία και το γεγονός ότι σήμερα και χτες οι κόπτες και οι μουσουλμάνοι ε, περπατούν χέρι-χέρι είναι αρκετή απόδειξη για το ότι θέλουν μια πραγματική δημοκρατία. Και ένα δεύτερο παράδειγμα που θα σας δώσω, για να μην φοβόμαστε να εκφραστούμε υπέρ της δημοκρατίας. Όλοι γνωρίζετε τον Μοχάμετ Μποαζίζη, αυτόν που στην ουσία ξεκίνησε την ε, ε, επανάσταση στην Τινησία μέσω της αυτοπυρπόλησής του. Στο φέρετρό του δεν υπήρχε η πράσινη σημαία του Ισλάμ, υπήρχε, ήταν καλυμμένο με την κόκκινη σημαία της Τινησίας. Δεν είναι Ισλαμικές οι επαναστάσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή, είναι επαναστάσεις για την ελευθερία. Εδώ και σχεδόν μια εβδομάδα Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώνονται στο Κάιρο. Τη στιγμή όπου γίνονται ταυτόχρονα διαδηλώσεις στην Ιορδανία, στην Ιεμένη, στη Συρία, στην Αλγερία. Σας ρωτώ κυρία Άστον, σας ζητώ κυρία Άστον, αλλάξτε την στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θέλω να μας πείτε εδώ σήμερα, σε αυτή την αίθουσα, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει 100% το λαό της Αιγύπτου και τις διεκδικήσεις του. Και θα θέλαμε επιτέλους ο Μουμπάρακ να ακούσει το λαό του και να απελευθερώσει μέσω της αποχώρησής του τη χώρα του για τη δημοκρατία και την ελευθερία. Εγώ αυτή την απάντηση θέλω να ακούσω στην, στην ομιλία σας. ο κύριος για 3,5 λεπτά. Ε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Άστον, κάνετε μια έκκληση στην ηρεμία αλλά θα πρέπει να πείτε τα πράγματα με το όνομά τους. Είναι τα προβλήματα του είναι ο Μουμπάγκ, ο οποίο εγκατέστησε τον τρόμο, την τρομοκρατία σήμερα στην Αίγυπτο. Δεν είναι οι διαδηλωτές. Λοιπόν, να μην ζητάτε να, να επικρατήσει ηρεμία. Ζητήστε από τον Μουμπάρακ να μην επιτεθεί στου ε, διαδηλωτέ, γιατί το κάνει για να πει στη συνέχεια ότι εγώ θα ξαναβάλω στο χάο σε τάξη. Αυτή είναι η παγίδα που μας στείνει και εμεί ε, να λέμε ότι θα πρέπει να επικρατήσει η ηρεμία. Όχι, να πούμε στο Μουμπάρακ να ηρεμήσει εκείνο. Και ο καλύτερο τρόπος να επικρατήσει η ηρεμία είναι να αποχωρήσει ο Μουμπάρακ και στην περίπτωση αυτή θα θριαμβεύσει, θα βασιλέψει η ηρεμία στο Κάιρο είδατε ότι ήταν οι αστυνομικοί του Μουμπάρακ αυτοί που έφτασαν με τα μαχαίρια. Ήταν φτωχοί από τα βάθη της Αιγύπτου που έφτασαν με λεωφορεία στην Αίγυπτο και δημιούργησαν τις ταραχές. Θα πρέπει να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους κυρία Άστον και να μην ε, προσποιούμεθα ότι είμαστε ε, τυφλοί. Και κάτι που βρίσκω εξ, ε, εντυπωσιακό. Σήμερα... Ε, όταν πριν από τρει εβδομάδε στην Τινησία εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, θέλαμε εμείς να πάρουμε μια πρωτοβουλία ζητώντας ε, να πάψουν οι διαπραγματεύσεις λόγω της δικτατορίας στην Τινησία μας λέγατε ότι αυτό δεν είναι δυνατό και σήμερα μας λέτε ξαφνικά ότι, είναι δυνατό είστε εκ των υστέρων μια επαναστάτρια σας ζητώ κυρία Άστον το εξή όσον αφορά την Τινησία να μας πείτε Πού έβαλε η Ευρώπη τα χρήματα, πείτε μας σε ποιες επιχειρήσεις ε, πήγαν τα ευρωπαϊκά χρήματα, τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Ποιε είναι οι επιχειρήσει του κυρίου Πεναλή και τη γυναίκα του που στηρίχθηκαν από τα ευρωπαϊκά, ευρωπαϊκά κονδύλια. Ε, μπορείτε να μα το πείτε, γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει το δικαίωμα να γνωρίζει, να ξέρει. Δεύτερον, κυρία Άστον, εφόσον λέτε ότι θέλετε να υποστηρίξετε σήμερα το λαό τη Τινησία, σα ρωτώ ένα πράγμα. Δηλαδή, ε, μετάβαση να υπάρχει μια ισότητα ευκαιριών στη δημοκρατική διαδικασία. Και αν γίνουν νέε εκλογέ, ξέρετε ότι το RCD έχει χρήματα και οι αντιπολιτευτικές δυνάμεις που ήταν απαγορευμένες επί χρόνια δεν διαθέτουν χρήματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θα πρέπει να πάει και να υποστηρίξει τη δημοκρατία και την ισότητα των όρων. Όσον αφορά τώρα την Αίγυπτο, κύριε Άστον, υπάρχει κάτι το οποίο είναι προφανές σήμερα εάν δεν ε, πετύχουμε να υποστηρίξουμε τους Αιγυπτίους, τον Αιγυπτικό λαό σε αυτή τη ε, διαδικασία απελευθέρωσης, τότε οι λαοί της Μέσης Ανατολής, οι αραβικοί λαοί, θα μας, ε, στρέψουν, θα μας γυρίσουν την πλάτη. Ενώ σήμερα έχουμε πραγματικά μια εξαιρετική κατάσταση μπροστά μας. Έγινε μια διαδήλωση στη Γάζα υποστήριξης προς τους Αιγυπτίους και η Χαμάς ε, απαγόρευσε την ε, ε, πάταξη της διαδήλωσης και αυτή είναι η απόδειξη ότι το πνεύμα, ο άνεμος της ελευθερίας στρέφεται κατά των θεοκρατικών καθεστώτων στη Μέση Ανατολή και στις αραβικές χώρες και είναι ο δικός μας ρόλος να τους υποστηρίξουμε. Ε, χύσαμε δάκρυα για επιχρόνια χρόνια λέγοντας ότι δεν υπάρχει καμία εναλλακτική δυνατότητα μεταξύ δικτατορίας και θεοκρατίας αλλά Ευτυχώς υπάρχει μια τρίτη δυνατότητα, η ελευθερία και η μάχη υπέρ της ελευθερίας κατά της θεοκρατίας και κατά της δεκτατορίας και ο ρόλος μας είναι να στηρίξουμε αυτούς που ηγούνται αυτού του αγώνα. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Άστον. Κύριε Βέλε, ε, σηκώσατε ένα, μια μπλε καρτέλα. Αυτό ήταν για να τραβήξει την προσοχή μου ή για να ρωτήσετε κάτι τον κύριο Κονμπεντίτ. Κύριε Κονμπεντίτ, δέχεστε ερώτηση από τον κύριο Βέλε. 30 δευτερόλεπτα έχετε. Hold on a second. Microphone. Μικρό λεπτό. Okay. I do. Okay. Go ahead. With all due respect to... Με όλο το σεβασμό στον κύριο Φερχόφστατ, και τον κύριο Κόνβεντιτ. Είστε πολύ διάσημο στη χώρα, χώρα σας. Συγγνώμη που δεν το λέω, δεν θυμάμαι εγώ το όνομά σας. κυρία Επίτροπε, εγώ έχω πολύ σοβαρές αντιρρήσεις για τα όσα είπαν οι δύο κύριοι. Αυτή όλη η κατάσταση θυμίζει το Ιράν. Παρακαλώ, προσοχή στο χειρισμό της Βορειοαφρικής. Δεν είναι η Ευρώπη η Βόρεια Αφρική. Το ερώτημά μου είναι, θυμάστε τι έγινε στο Ιράν. Δεν βλέπετε καμιά ομοιότητα. Δεν συμφωνείτε ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε μια τακτική μετάβαση. Εκτός μικροφώνου η δεν τολμώ εγώ να σας κάνω βέβαια μάθημα ιστορίας. Να σας θυμίσω όμως ότι στο Ιράν η Δύση, η Αμερική στήριξε τον Σάχη. Και μέχρι την τελευταία στιγμή ακόμα και με υπό την κυβέρνηση Μπαξιά, εμείς ήμασταν στη λάθος πλευρά. Και ότι δώσαμε όλα τα όπλα στη θεοκρατία του Ιράν για να κερδίσει. Αυτό ήθελα να σας εξηγήσω, ότι αν δεν είμαστε από την πλευρά των όσων αγωνίζονται για την ελευθερία, αυτοί που αγωνίζονται για την ελευθερία θα βρεθούν σε αδιέξοδο και η άλλη πλευρά είναι αυτή που θα κερδίσει. Αυτό ακριβώς είναι το δίδαγμα του Ιράν. Το Ιράν είναι αυτό που είπε ο κύριος Γρομπατσόφ, που όποιο στάσει πολύ αργά στην ιστορία θα χάσει. Για μια φορά λοιπόν η Ευρώπη να μην φτάσει καθυστερή εξερημένα στην περιοχή. Εξ ονόματος των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών, ο κύριος Τάνοκ για δύο λεπτά σε ένα άλλο θέμα τώρα δεν θα μιλήσω για το ποιοι οδήγησαν τον Χομέινι στον Τεχιράν. Λοιπόν, ο Μουμπάρακ είναι ο τρίτος πρόεδρος της συγκεκριμένης χώρας, την, την Ισία. Ο Μπεναλή ήταν ο δεύτερος ηγέτης μετά από την ανεξαρτησία. Όταν τέτοιου είδους κινήσεις οδηγούν σε βίες αλλαγές βλέπουμε ότι είναι ανεξέλεκτα τα πράγματα. Τώρα υπάρχει μια καταιγίδα αλλαγών. Η πολιτική μου ομάδα ζητά να υπάρξει μια μετάβαση ειρηνική και δημοκρατική. Ενώ σήμερα είδαμε ότι υπάρχει μια στροφή ανησυχητική στη βία. Ε, δεν μπορούμε να καταλάβουμε ε, κάποιον τρόπο να συνεισφέρει στη μετάβαση αυτή ο Μουμπάρακ εκτός από το να παρετηθεί. Νομίζω ότι και στην Τινησία ε, το καθεστώς ήταν μεν απολυταρχικό και διεφθαρμένο αλλά παρόλα αυτά παρήχε ένα ποσοστό ελευθεριών. Και αυτή τη στιγμή στην Αίγυπτο οι αδελφοί μουσουλμάνοι προσπαθούν να καλύψουν το λεγόμενο πολιτικό κενό το οποίο είχε δημιουργηθεί στη χώρα αυτή. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα και στις σχέσεις τους με τις γειτονικές χώρες όπως επίσης και στη λειτουργία της σύραγγας του Σουέζ, της διορία συγγνώμη του το να υπάρξει μια φιλελεύθερη δημοκρατία χωρίς καμία παράδοση σε αυτές τις χώρες, οι Ηνωμένε Πολιτείε, η Ευρωπαϊκή Ένωση και όλοι οι πολιτικοί ε, ε, σκεπτόμενοι άνθρωποι πρέπει να βοηθήσουν και να στηρίξουν αυτούς οι οποίοι θα υποστηρίξουν στις χώρες αυτές ε, την πολιτική ελευθερία και θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουμε κινήσεις όπως αυτές τις οποίες θα κάνουν προετοιμαζόμενοι για τις επόμενες εκλογές οι αδελφοί μουσουλμάνοι. Θα λειτουργήσει ε, θα έλεγα σαν υπόδειγμα αυτό το οποίο θα γίνει στην Αίγυπτο και στις άλλες χώρες. Υπάρχουν και άλλα παραδείγματα στην Ινδονησία σαν παράδειγμα και στην Τουρκία για μουσουλμανικά καθεστώτα τα οποία λειτουργούν με δημοκρατία και μπορούν να πάρουν παραδείγματα από τις χώρες αυτές η Αίγυπτος και η Τινησία που θα οδηγήσει στη σταθερή και διαρκή δημοκρατία. Ο κύριος Μπέλα, μπλε κάρτα. Κύριε Τάνοκ, δέχεστε την ερώτηση. Θα ήθελα να πω στον κύριο Τάνοκ ότι η στάση του σε σχέση με αυτούς οι οποίοι έχουν εξεγερθεί σήμερα είναι απαράδεκτη. Η εξέγερση είναι μια λαϊκή εξέγερση και ο λαός στις χώρες αυτές ζει σε μια, σε μια απέραντη φτώχεια και γι' αυτό έχει εξεγερθεί σήμερα και οι δικτάτορες που κυριαρχούσαν στις χώρες αυτές υποτίθεται ότι για να αποτρέψουν τον Ισλαμισμό ε, καταπιέζουν τον κόσμο. Εσείς λοιπόν να μας πείτε ο λαός στις χώρες αυτές έχει το δικαίωμα εξέγευσης ή όχι. Κοιτάξτε τα διευκρίνησα αυτά λέει ο κύριος ε, Τάνο και εγώ δεν θέλω σε καμία περίπτωση ο Χωμεϊνή ή οποιοδήποτε άλλος θεοκράτης να κυριαρχήσει στις χώρες αυτές. Προτιμώ με ελεύθερες εκλογές να βγει ένας δημοκράτης που θα κυριαρχήσει στις χώρες αυτές και τα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα στις δύο χώρες είναι τεράστια. Δεν είναι αυτό όμως το θέμα σε αυτή τη φάση. Σε αυτή τη φάση είναι να διασφαλίσουμε μια διατεταγμένη και ειρηνική μετάβαση και όχι μια κατάρρευση της τάξης στις χώρες αυτές. Γιατί εμείς θέλουμε την ειρήνη στην γειτονία μας. Ίσως θα πρέπει να σας δώσουν κάποιες εξηγήσει οι φιλελεύθεροι δημοκράτες, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της ομιλίας σας φάνηκε να διασκεδάζουν. Κυρία Βερζιά. Oui, merci. Ε, ε, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δεν ήθελα τόσο να επανέλθω στο παρελθόν, αλλά ακούω κάποιες εντυπωσιακέ παρεμβάσεις. Βρίσκω ότι τελευταία επί μήνες είμαστε κάπως απομονωμένοι με κάποιους πράσινους βουλευτές για να ζητήσουμε να γίνει συζήτηση για την κατάσταση στην ε, Ισία. Ε, πράγματι, κύριε Κονμπετίτ, έχετε δίκιο. Υπάρχουν ε, πολλοί επαναστάτες της ίστατης στιγμής, εκ των υστέρων. Ε, είπαμε κάποια πράγματα στο ίδιο μας το ψήφισμα και νομίζω ότι θα πρέπει να στρέψουμε τα μάτια μας προς το παρελθόν αλλά στο μέλλον. Θα πρέπει να, να αποφύγουμε κάθε παρέμβαση στα εσωτερικά αυτής της χώρας. Δεν αναπόκειται σε εμάς τους Ευρωπαίους να πούμε πώς οι κυβερνήσεις αυτής της χώρας θα πρέπει να ε, σχηματιστούν. Ο λαός της ε, Τινησία απελευθερώθηκε μόνο του το δικτατορικό, από το δικτατορικό καθεστώ. Α εκφραστεί μόνο του ο λαό και α υποστηρίξουμε τη μετάβασή του προ τη δημοκρατία. Όλοι όσοι παρακολουθούν την κατάσταση στην Ισία γνωρίζουν ότι το παρελθόν δεν έχει ακόμη πεθάνει και ορισμένοι κάνουν κάποιου ελιγμού και χειραγούν τα πράγματα στη σκιά. Η βία σήμερα στην Τινησία δείχνει πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Ναι, να καταδικάσουμε στεναρά κάθε μορφή βία. και μην αρκείστε να ζητάτε απλώς να συγκρατηθεί η βία όπως κάνατε για την Τινησία. Ε, η αστυνομική βία είναι απαράδεκτο στην Ισία, στην Αίγυπτο και σε όλες τις περιοχές του κόσμου. Ζητήσουμε από τις αρχές της Ισίας και το λαό της Ισίας αυτό το οποίο αναμένουν από εμά χωρίς να θέλουμε να τους επιβάλλουμε τίποτα. Ε, κάνατε κάποιες ε, συζητήσεις αλλά προσθέσατε ότι θέλετε να αυξηθεί η πρόσβαση στις, αγοράς, στις αγορές. Θεωρώ ότι αυτό είναι άστοχο. Όλοι μοιάζουν να ανακαλύπτουν σήμερα την διαφθορά του καθεστώς του κυρίου Μπαναλή. Η, απελευθέρωση στην, ε, η οικονομική απελευθέρωση στην Ισία ήταν εις του Μπαναλή και της οικογένειάς του χάρη στην βοήθεια των Ευρωπαίων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχασε μεγάλο βαθμό αξιοπιστία σε αυτή τη χώρα, όπου θα πρέπει επιτέλους να υποστηρίξουμε τους δημοκράτες και να καταδικάσουμε όλες τις δικτατορίες. κύριος Προβέρα για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η παλαιά πολιτική τάξη στο Μαγκρέμπ καταραίει και δημιουργούνται πάρα πολλά νέα προβλήματα από την κρίση αυτή. Μαζί με τις ελπίδες υπάρχουν και οι κίνδυνοι. Υπάρχει περίπτωση κάποια, θεο... κάποια καθεστώτα τα οποία ήταν φυσικά μη θρησκευτικά και όχι δημοκρατικά να αντικατασταθούν από θεοκρατικά καθεστώτα αντιδημοκρατικά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να συνοδεύσει κανείς με δημοκρατικό τρόπο μια εξέγερση και μια επανάσταση και από το Ιράν θα πρέπει να βγάλουμε κάποια μαθήματα, θα έλεγα, κάποια συμπεράσματα. Η κρίση φοβάμαι ότι θα χειροτερεύσει τα προβλήματα την ανεργία των νέων και τις μεταναστευτικές ροές τις οποίες δεν μπορεί να αντέξει η Ευρώπη. Τα γεγονότα αυτά αντιπροσωπεύουν και την ανεπάρκεια της ευρωμεσογειακής πολιτικής και την πολιτική συνεργασίας που είχαμε με τις χώρες αυτές μέχρι τώρα που είναι ανεπαρκής για να δημιουργήσει συνθήκες ανάπτυξης και δημοκρατίας. Αυτά τα οποία συνέβησαν δεν οφείλονται μόνο στην οικονομική κρίση αλλά και στην έλλειψη κοινωνικής συνοχής και σταθερότητας, στην έλλειψη εκπροσώπησης των λαϊκών συμφερόντων, στην έλλειψη συνδικάτων ελεύθερου τύπου, πλουραλισμού των κομμάτων του τύπου του κράτους δικαίου και των ισότιμων ευκαιριών για όλους. Το να συνοδεύσουμε τις χώρες αυτές στις νέες διαδικασίες πρέπει να είναι ο βασικός στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μαζί με την οικονομική συνδρομή. Τότε θα δημιουργήσουμε την πραγματική σταθερότητα, τη σταθερότητα ενός όχι θεοκρατικού καθεστώτος, αλλά ενός καθεστώτος που βασίζεται στους δημοκρατικούς θεσμούς και στη συμμετοχή. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν, κατά την άποψή μου, καθώς ε, ετοιμάζομαι για αύριο για την ad hoc αποστολή στην Τινησία, το θέμα είναι να στηρίξουμε το λαό της Τινησίας και να θυμόμαστε πόσο σημαντικό είναι και ενώ σεβόμαστε τις πολιτιστικές του αξίες και την ταυτότητά τους, να τους βοηθήσουμε να φτιάξουν ένα νέο μέλλον με βάση το κράτος δικαίου και τα δημοκρατικά ιδανικά. Ο κόσμος περιμένει αλλαγή και βοήθεια χωρίς ε, περιορισμούς. Εγώ είμαι πολύ ευτυχής που ο κύριος Κον Μπεντίτ ακολούθησε αυτό που είπα εγώ στην αντιπροσωπή σήμερα το πρωί σε σχέση με το ακριβώς τι συνέβη με τα χρήματα τη Ένωση όλα αυτά τα χρόνια. Ο εκπρόσωπος της ΕΕΣ ε, είπε ότι δαπανήθηκαν σε μεταρρυθμίσεις. Μα τι είναι μεταρρυθμίσεις. Άμα είχαν γίνει μεταρρυθμίσεις ο κόσμος δεν θα είχε επαναστατήσει με τον τρόπο που επαναστάτησε. Χρειάζεται να οθήσουμε την προσωρινή κυβέρνηση, να διερευνήσει πού πήγαν αυτά τα λεφτά και να εξασφαλίσουμε ότι οποιαδήποτε χρήματα σταλούν στο μέλλον να δαπανώνται και σωστά. Ε, ο ο αραβικός κόσμος είναι ο εταίρε μας στην Ένωση για τη Μεσόγειο. Σε, όλη μας ε, σε όλες μας τις επαφές μαζί τους πάντοτε προτείναμε ε, τις ε, αρχές του πλουραλισμού, της δημοκρατίας, της ελευθεροτυπίας, ε, της ελεύθερης συγκέντρωσης, της ανεξαρτησίας και της χρηστής διαχείρισης. Και ανέκαθεν υποστηρίζαμε ότι όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν από το εσωτερικό και να μην επιβληθούν από ε, ε, άλλους εκτός των χωρών αυτών. Ο λαός της Τουνησίας κατάφερε εκ των έσω να ε, να διώξει την καταπίεση και το απολυτερχικό καθεστώ. Θα πρέπει λοιπόν οι τρισικέ αρχέ να σεβαστούν τη βούληση του λαού και να προχωρήσουν χωρί καθυστέρηση στη διαδικασία εκδημοκρατισμού και λογοδοσία σε περιπτώσει διαφθορά ή καταπίεση ή καταστολή από τους ε, παρατρεχάμενους του Μπεναλή. Για τους ίδιους λόγους, ε, ο λαός της Αιγυπτίου έχει ψηφίσει τα συλλήψεις, ε, τις δολοφονίες ε, και απέτησε την ελευθερία και την ε, χειραφέτηση. Ελευθερία δεν σημαίνει μόνο εκλογές σημαίνει και δημοκρατία δεν σημαίνει μόνο εκλογές, σημαίνει πολύ περισσότερο από αυτό. Εμείς ανεπιφύλακτα υποστηρίζουμε το λαό της Αιγύπτου και καλούμε τους σημερινούς του ηγέτες να ακούσουν την σοφία του λαού τους και να μην αποτελέσουν εμπόδιο στην ανταπόκριση στις προσδοκίες τους στους δικούς μας Ευρωπα... Ευρωπαίους υπαλλήλους, στο Συμβούλιο και το ενίπατο το εκπρόσωπο εγώ θα πω το εξής. Είναι απογοητευτικό να ακούει κανείς τον πρόεδρο Ομπάμα ή τη Χίλαρη Κλίντον να μιλούν τολμηρά και εγκαίρως και εσείς όπως πάντα να παίζετε το δεύτερο βιολί. Και αυτό ίσα ίσα που να ακούγεται. Κυρία Ντεκάιζερ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Υπάρχουν πράγματι κάποιες στιγμές όπου θα πρέπει κανείς να ξέρει να διαλέξει στρατόπεδο. Και το στρατόπεδο σήμερα είναι απολύτως ξεκάθαρο. Είναι ξεκάθαρο, το είπαν άλλωστε και οι συνάδελφοι, είναι η οδός προς την ελευθερία, είναι η οδός του λαού. Λοιπόν, τη στιγμή που σας μιλώ, το Μουσείο του Καΐρου φλέγεται, οι μάχες ξεσπούν στους δρόμους και πιστεύω ότι για την Αίγυπτο, εν πάση περιπτώσει, πραγματικά δεν υπήρξαμε αρκετά ξεκάθαροι. Ο Μουμπάρακ θα πρέπει να φύγει, αυτό είναι ξεκάθαρο. Ο Μουμπάρακ, όπως είναι και πραγματικά σέβομαι τον παλιό του αγώνα. Ο Μουμπάρακ όπω είναι δεν είναι σε θέση να ολοκληρώσει τη δημοκρατική μετάβαση. Είναι τρέλα να ζητάει κανεί κάτι τέτοιο και να αφήνει ε, το στατόπεδο, τους οπαδούς του Μουμπάρακ ε, στους δρόμους του Καϊούρ ελεύθερους να έρχονται σε ψημαχίες με τους ε, ε, οπαδούς της αντιπολίτευσης εγώ διερωτήθηκα κατ' επανάληψη ποια είναι τα σφάλματα που κάναμε και κάναμε ένα μείζον σφάλμα. Το σφάλμα ήταν να υποστηρίζουμε διεφθαρμένα καθεστώτα εις το όνομα της σταθερότητας χωρίς να λαμβάνουμε καθόλου υπόψη μας το ζήτημα της κοινωνικής δικαιοσύνης και την ε, βούληση ελευθερίας του λαού. Το δεύτερο σφάλμα, και λυπούμε αγαπητοί συνάδελφε, είναι ότι δεν κατανοήσαμε το πολιτικό Ισλάμ. Δεν λέω ότι δεν αποδεχθήκαμε το πολιτικό Ισλάμ, γιατί υπάρχει μια διαφορά μεταξύ της θερμοκρατίας των φονταμενταλιστών και, ορισμένων αδελφών, και των αδελφών μουσουλμάνων. Ε, θα πρέπει να κάνουμε αυτή τη διάκριση. Γιατί εμείς σήμερα εκθρέψαμε το φονταμενταλισμό, εκθρέψαμε ε, την τρομοκρατία. Και ε, επίσης θα πρέπει να διατηρήσουμε τα κεκτημένα του παρελθόντος της Αιγύπτου και της ε, Τινησίας, δηλαδή τις κοσμικές δομές του κράτους, τα δικαιώματα των γυναικών που είναι σημαντικά σε αυτές τις χώρες. Συνεπώς λοιπόν τις λαϊκές κοσμικές δομές αυτών των κρατών, να απομακρύνουμε τον Ισλαμικό νόμο. Ε, μπορούμε να στηρίξουμε τη δημοκρατική μετάβαση διαφυλάτοντας αυτή την ιδέα του κοσμικού χαρακτήρα, του λαϊκού χαρακτήρα του κράτους, σεβόμενη την θρησκευτική πίστη και τις διαφορές μεταξύ των λαών, τις πίστη και τις διαφορές. Thank you, um, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω πως σήμερα το κατεπήγον θέμα είναι η κατάσταση στην Αίγυπτο. Το 2005 ήμουν πρόεδρο μια ε, μικρή ε, αποστολή παρατηρητών για τι εκλογέ εκεί. μα ζητήθηκε να πάμε για τον πρώτο γύρο και για το δεύτερο γύρο. Αλλά ο πρώτο γύρο ήταν τόσο χαοτικός και τόσο χάλια, τόσο διεφθαρμένο που αποφασίσαμε να μην πάμε καν στο δεύτερο γύρο. Είναι μια χώρα η Αίγυπτος όπου για 30 χρόνια ένας δικτάτορας, ο Μουμπάρακ, έχει συγκεντρώσει απόλυτη εξουσία σε ένα βίο καθεστώς και αν και όλοι αναγνωρίζουμε την ε, φοβερή ε, εξέλιξη στους δρόμους της Αιγύπτου, βλέπουμε ότι ο Μουμπάρακ αντιδρά σαν κάποιος που ξέρει ότι υποστηρίζεται όχι μόνο από την Αίγυπτο μέσα, αλλά και αλλού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση γνωρίζει ότι μπορεί μόνο ηθική, ηθικό κύρος να ε, δείξει. Όταν η Βαρόνη Άστον ε, μίλησε έτσι διστακτικά στην αρχή, ξέρει ότι δεν έχει και μεγάλες, ε, μεγάλη δυνατότητα πειθούς. Θα πρέπει ωστόσο να μιλάμε με μια φωνή τουλάχιστον. Και δεν έχουμε μιλήσει με μια φωνή μέχρι στιγμή. Αναφέρθηκε προηγουμένω. Οι πρωθυπουργοί τη ε, Γαλλία, τη ε, Αγγλία, τη Μεγάλη Βρετανία και τη Γερμανία μίλησαν χώρια. Θα πρέπει να ξέρουμε πού βρισκόμαστε, να στηρίζουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο και ειδικά αυτή τη στιγμή για τη Μεσόγειο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Άστον. Θα ήθελα να επαναλάβω την έκκληση κυρία Άστον ε, να μας πείτε που πήγαν τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί υπάρχουν κάποιοι φόβοι ότι η οικογένεια του Μπεναλή επωφελήθηκε από αυτά τα κονδύλια. Ε, νομίζω ότι χρειάζεται μια ξεκάθαρη ανακατανομή των κονδυλίων ε, και στην Τινησία χρειαζόμαστε έναν καινούριο επικεφαλή τη αντιπροσωπεία. Θα ήθελα να σα διαβάσω ότι έγραψε σήμερα σε ένα email. Η ευρωπαϊκή στρατηγική στην Τινησία δεν χρειάζεται να αναθεωρηθεί. Θα υπάρχουν περισσότερε ελευθερίε στι επιλογέ μα, αλλά ε, οι συμφωνίες μας ε, έχουν ακόμα μεγαλύτερη σημασία σήμερα. Θεωρώ ότι είναι ε, απίστευτο αυτό το οποίο γράφετε, ότι δηλαδή θα πρέπει να αναθεωρηθεί η δική μας πολιτική εναντί της Τινησίας και σας καλώ να αναλάβετε πρωτοβουλία να αλλάξει ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας. Και θα ήθελα να προσθέσω ένα σημείο σε σχέση με τα όσα ανέφερε η κυρία Κάιζερ. Νομίζω ότι είναι καιρός να υποστηριχθούν οι γυναίκες σε αυτή τη μεταβατική φάση. Γιατί τι δεν κάνετε μια συνδιάσκεψη με την δική σα υποστήριξη εκεί ε, για τις ε, γυναίκες σε αυτή τη μεταβατική φάση για να φωτίσετε το ρόλο του και να τις στηρίξετε ούτως ώστε να τονίσετε τον κοσμικό χαρακτήρα αυτής της δημοκρατικής μετάβασης της χώρας αυτές. Νομίζω ότι αυτό θα έχει προτεραιότητα σε μια τέτοιου είδου ατζέντα. Ευχαριστώ πολύ. Οι μαζικές διαμαρτυρίες στην Ισραήλ και στην Αίγυπτο στην στρατηγική σημασία Αίγυπτο έχουν ε, ε, προκαλέσει την προσοχή όλων των δυνάμεων σε ολόκληρο τον κόσμο. Υπάρχουν διάφορα σενάρια. Η ειρηνική ανάληψη της εξουσίας από τις προοδευτικές δυνάμεις, αλλά και ακόμα και εμφύλιος, χωρίς να αποκλείται και το, η περίπτωση της χρήσης πυρηνικών όπλων. Είναι ιδιαίτερα ε, ευαίσθητη η κατάσταση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να κρατήσει, να να κρατήσει κοινή στάση και να ε, υποστηρίξει τη σταθεροποίηση στην περιοχή. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε το ψήφισμα που υιοθετήσαμε πρόσφατα για τη δίωξη χριστιανών που ίσχυε και για την Αίγυπτο. Θα πρέπει λοιπόν να προβούμε σε συγκεκριμένα βήματα και να στείλουμε αποστολή παρατηρητών στην Αίγυπτο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρία Άστον. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αναθεωρήσει την πολιτική γειτονία τη. Γιατί είναι αλήθεια κυρία Άστον ότι δίνουμε την εντύπωση ότι μα ανησυχούν περισσότερο οι συμφωνίε ελεύθερου εμπορίου παρά η εξέλιξη των λαών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το πρόβλημα, κυρία Άστον, δεν είναι τόσο η θέση που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με το καθεστώ του Μπεναλή και του Μουμπάρακ, αλλά ποια είναι η θέση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, σε σχέση με το παρελθόν και σε σχέση με τις αλλαγές που ζήτησαν οι πολίτες στους δρόμους. Αυτό είναι το πρόβλημα που καλείται να επιλύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ότι δεν δηλώνουμε τη δική μας παρουσία στις αλλαγές που ζητούν οι λαοί όχι μόνο της Τινησίας αλλά του Μαρόκο, της Αιγύπτου, της Ιορδανίας, της Ιεμένης και πραγματικά πάρα πολλοί λαοί οι οποίοι δεν αντέχουν πλέον τα αυταρχικά καθεστώτα και μια κρίση η οποία καταφέρει κέριο πλήγμα στους πιο αδύναμους. Αυτή είναι η ενθόρυση που πρέπει να κάνει με τα ρύθμιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να αλλάξει την, ριζικά την πολιτική γειτονία της. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν εκπλήσεται κανείς από το ότι τα γεγονότα στην Τινησία και ιδιαίτερα στην Αίγυπτο προκαλούν τεράστιο ενδιαφέρον σε όλες τις χώρες αλλά ιδιαίτερα στο Ιράν. Έχει ενδιαφέρον λοιπόν να προσπαθήσει κανείς να κατανοήσει την στάση ε, της Ιρανικής κυβέρνησης η οποία χαιρετίζει ε, την άφηξη του επαναστατικού κύματος και στην Αίγυπτο. Φαίνεται λοιπόν ότι προσπαθούν να καλύψουν οι Ιρανοί θεοκράτες τις εξεγεύσεις στις δύο αυτές χώρες και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να υποτιμήσει τον κίνδυνο μιας ριζοσπαστικοποίησης του αραβικού κόσμου. θα πρέπει αυτή η εξέγερση να μην χρησιμοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο που χρησιμοποιήθηκε η αντίστοιχη στο Ιράν. Κύριε Πρόεδρε, αυτά τα οποία συμβαίνουν σήμερα στην Τινησία και την Αίγυπτο έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία έχουν εξεγερθεί οι κάτοικοι των χωρών αυτών εναντίον των δεσποτικών παλαιών καθεστώτων. Το θέμα είναι τι θα αντικαταστήσει αυτές τις δικτατορίες πλέον. Αυτό είναι και το παράδοξο αν θέλετε του εκδημοκρατισμού στις μουσουλμανικές χώρες. Η περισσότερη δημοκρατία πολλές φορές επιτρέπει την μεγαλύτερη παρουσία φυσικά και των Ισλαμιστών και αυτό δημιουργεί ορισμένα διλήμματα. Θα πρέπει λοιπόν η εξουσία να πέσει στα χέρια των πραγματικών δημοκρατών. Δεν ξέρω τι ρόλο θα μπορούσαν να παίξουν ε, οι αδελφοί μουσουλμάνοι, γιατί αν δημιουργηθεί ένα θεοκρατικό καθεστώς στην Αίγυπτο, τότε θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε καταστάσεις αντίστοιχες με αυτές του Ιράν. Ας είμαστε λοιπόν πάρα πολύ προσεκτικοί. Θυμίζω ότι μέχρι πριν λίγες εβδομάδες ο Μπεναλή και οι φίλοι του ήταν μέλη της Σοσιαλιστικής Διεθνούς. Λοιπόν, ας μην ξανακάνουμε τα ίδια λάθη, ας είμαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί στην επιλογή των φίλων μας των πολιτικών. Η κυρία Σίνκλερ, ζητήσατε το λόγο. Όχι. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Ήπατη, εκπρόσωπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η δική μας απάντηση στα τεκτενόμενα στον αραβικό κόσμο θα πρέπει να προκύπτει από την εικόνα μας για τον άνθρωπο, την κοσμοθερία μας. Ο κάθε άνθρωπος, είτε είναι χριστιανός, αμαμεθανός, εβραίος ή άθεος, έχει το ίδιο δικαίωμα αξιοπρέπειας και το ίδιο δικαίωμα να ζει σε αξιοπρεπείς συνθήκες. Και από αυτό προκύπτει και από, εδώ, από εκεί προκύπτει το δικαίωμα των λαών αυτών να ζουν σε συνθήκες ελευθερίας, δημοκρατίας και σε ένα καθεστώς το οποίο σέβεται την ανθρώπινη εξωπρέπεια. Γι' αυτό σήμερα είναι το καθήκον μας, η ευθύνη μας και ε, το σημαντικότερο μέλημά μας για το μέλλον να στηρίξουμε τους ανθρώπους στον αραβικό κόσμο που μάχονται ειρηνικά για την ελευθερία και τη δημοκρατία και να τους πούμε ότι στεκόμαστε αλληλέγγυοι στο πλευρό τους, είμαστε αλληλέγγυοι με τους ειρηνικούς μου αμεθανούς ε, στον αραβικό κόσμο. Αγαπητοί συνάδελφοι, διαπράξαμε μια φορά το σφάλμα σε σχέση με τον ε, ολοκληρωτικό κομμουνισμό να κλείσουμε τα μάτια γιατί είπαμε ότι χρειαζόμαστε σταθερότητα. Αυτό το σφάλμα δεν θα πρέπει να επαναλάβουμε σήμερα, γιατί στη σταθερότητα ανήκει, συμπεριλαμβάνεται η ελευθερία και η δημοκρατία και θα πρέπει να το υποστηρίξουμε. Και όταν ακούμε εδώ αυτές τις στιγμές ε, δεν ήξερα ότι πέφτουν πυροβολισμοί στο Κάιρο και μέχρι τώρα ο στρατός τόσο στην Τινησία όσο και στην Αίγυπτο ήταν συγκρατημένο. Εάν ο στρατός προσπαθήσει να επιβληθεί με τη βία ε, αυτό δεν μπορεί παρά να κρατήσει ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Στην Ευρώπη το 1953 είχαμε την Επανάσταση στην Ανατολική Γερμανία, το 1956 στην Ουγγαρία, το 1968 στην Τσεχοσλοβακία και στη συνέχεια ήρθε η, Σολιτα... η ε, ε, θα πρέπει λοιπόν να πούμε δυνατά ας πάψουν οι πυροβολισμοί και δώστε στους ανθρώπους την ελευθερία να εκλέξουν το καθεστώς που επιθυμούν ειρηνικά. Και θα πρέπει να το υποστηρίξουμε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Υπάτη εκπρόσωπο, υπάρχουν κάποιοι οποίοι λένε ότι δεν μπορούμε να αντιλήσουμε διδάγματα από την ιστορία. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι θα πρέπει να το προστασίσουμε Και όταν αναφέρεστε κυρία Τζαβέλα στο Ιράν και ο κύριος Κονμπεντίτ σας έδωσε κάποια απάντηση, θα ήθελα να σας επισημάνω τι έγινε τότε στο Ιράν. Ε, πραγματικά στηρίξαμε ένα βρώμικο καθεστώς. Ε, στηρίξαμε το, την αστυνομία, ή ανεχθήκαμε την αστυνομία της χώρας αυτής που έκανε βασανιστήρια στους πολίτες. Και η Αμερική και η Μεγάλη Βρετανία ε, ε, ε υποστήριξαν μια ειρηνική ε, πανάσταση. Εμείς είμαστε πιο πίσω. Και ε, θα πρέπει να πω ότι συμφωνώ με τον συνάδελφο κύριο ε, Κονμπεντίτ. Θα πρέπει να σταθούμε στο πλευρό εκείνων που προώθησαν αυτή την επανάσταση που την ξεκίνησαν. Και δεν ήταν οι Ισλαμιστέ, α χαιρόμαστε για αυτή τη μεγάλη ευκαιρία που έχουμε ότι η επανάσταση δεν προήρθε από του Ισλαμιστέ, αλλά από του ανθρώπου στον δρόμο, από του πολίτε οι οποίοι δεν ήταν ικανοποιημένοι ούτε με την οικονομική κατάσταση ούτε με το δημοκρατικό έλλειμμα. Αυτό, αυτή είναι η κατάσταση που επικρατούσε τότε εκεί. Και αγαπητοί ε, συνάδελφοι, ας ασκήσουμε κριτική στους αυτούς μας. Ε, έχει καταρρεύσει ένα κομμάτι της πολιτικής μας γειτονίας, η οποία στηρίχτηκε στην επιθυμία να υπάρχει σταθερότητα και ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Θεωρήσαμε ότι η ειρήνη στη Μέση Ανατολή πρέπει να στηριχθεί στις πλάτες των δικτατόρων. Αυτό δεν είναι δυνατόν Γι' αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει να μιλήσουμε καθαρά, ξεκάθαρα. Ε, Στα δυνακές η ειρήνη στη Μέση Ανατολή μπορεί να εμπεδοθεί εφόσον εδράζεται στην ειρήνη και όχι στι δικτατορίε. Ε, κυρία Υπάτη, εκπρόσωπε, θα πρέπει να πούμε δυνατά ε, τη γνώμη μας. Ε, θα πρέπει να μιλήσουμε τόσο ηχηρά ότι ώστε να εισακωστούν οι, η, φωνή μας, η φωνή της Κάθριν Άστον και όχι της Χίλαρη ε, Κλίντον. Αυτό αναμένουμε από εσά να μιλήσετε μια ξεκάθαρη και δυνατή γλώσσα. λεπτό. Благодаря, господин председател, уважаема госпожо Остин, уважаеми колеги. Ευχαριστώ ε, κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμη κυρία Άστον, αγαπητοί συνάδελφοι. Οι διαμαρτυρίες στην Αίγυπτο κατά της κοινωνικής αδικίας, κατά της βίας και της ε, διαφθοράς στο σώμα της αστυνομίας, κατά των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δείχνουν ξεκάθαρα ότι οι άνθρωποι επιθυμούν μια αλλαγή και αυτό μας ε, θυμίζει την ε, κατάρρευση στις σοσιαλιστικές χώρες του Ανατολικού Μπλοκ. Το 89. Τα, το αίτημα του λαού, των λαών στην Αίγυπτο και στην Τινησία, ε, τα αιτήματα είναι απολύτως ξεκάθαρα. Θα πρέπει να στηρίξουμε αυτά τα αιτήματα γιατί επιθυμούν τον πλουραλισμό, επιθυμούν την ελευθερία του τύπου και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και γι' αυτό θα πρέπει, αγαπητή κυρία Άστον, να αναθεωρήσουμε την εξωτερική μας πολιτική στη βάση των αξιών μας θα πρέπει να χαράξουμε το δρόμο προς την δημοκρατία και να την υποστηρίξουμε. Θα πρέπει να ανταποκριθούμε στις επιθυμίες των ανθρώπων στην Τινησία και στην Αίγυπτο προκειμένου να χαράξουμε αυτό το δρόμο. Πρόεδρε, πριν από 60 χρόνια η επανάσταση στον αραβικό κόσμο σήμαινε απελευθέρωση από την ευρωπαϊκή Απικιοκρατία. 60 χρόνια μετά η επανάσταση σημαίνει αποκατάσταση της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Εμείς θα πρέπει να αποφασίσουμε με ποια πλευρά να σταθούμε. Το διακύβευμα είναι μια, μια ανεξάρτητη κοινωνία των πολιτών. Ε, ο δε προπολογισμό μας θα πρέπει να αναθεωρηθεί για να βοηθήσουμε την που έχει υποφέρει από 23 χρόνια από λιταρχικού καθεστώτος. Η πλειοψηφία αυτή ε, των νησίων δεν εμπιστεύονται την μη εκλεγμένη προσωρινή κυβέρνηση, υπηρεσιακή κυβέρνηση. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι πως η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μια πραγματική διαδικασία. Ήταν ε, τόσο μεγάλη η παραμέληση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας για τον αραβικό κόσμο όλα αυτά τα χρόνια. Και πραγματικά είναι αυτή η στιγμή για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Πρόεδρε. Thank you, Mr. Chairman. I do not share... Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ δεν συμμερίζομαι την άποψη ότι μια συνεχιζόμενη αναταραχή στην Αίγυπτο καθοδηγείται μόνο από δημοκρατικές δυνάμεις ευρωπαϊκού τύπου. Εγώ νομίζω αυτή, ότι αυτή η υποτιθέμενη επανάσταση για την αλλαγή κινητοποιείται ναι, για καλύτερη ζωή, αλλά το κρίσιμο ερώτημα για μας είναι, για μας τους Ευρωπαίους είναι η απειλή αυτή η δραματική κατάσταση να χειραγωγηθεί από ριζοσπαστικούς Ισλαμιστές. Αν γινόταν κάτι τέτοιο η Ευρώπη όπως και η Αμερική θα χάσει ε, ένα μετριοπαθή αραβικό, άραβα σύμμαχο και η Αίγυπτος θα μετατρεπόταν σε μια εχθρική χώρα που θα ερχόταν πιο κοντά στην Χαμάς. Η θέση της Ένωσης θα πρέπει να μείνει σταθερά στο πλευρό εκείνων που αναζητούν την ελευθερία και που, ε, και να υποστηρίξουμε ελεύθερες εκλογές. για ένα λεπτό. Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι φανερό ότι εδώ η συντριπτική πλειοψηφία του Κοινοβουλίου υποστηρίζει την εξέγερση των Αιγυπτίων. Και αυτό είναι πάρα πολύ σωστό, πλην βέβαια ελαχίστων εξαιρέσεων όπως αυτή που ακούσαμε μόλις τώρα. Όμω νομίζω και θα πρέπει να συμφωνήσετε μαζί μου ότι πολιτική σημαίνει να είναι κανεί έγκαιρος και κέριο και νομίζω ότι όλοι εμείς εδώ θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι δεν είδαμε αυτό που συνέβαινε στην Αίγυπτο αυτές τις τελευταίες δεκαετίες που ήμασταν εμείς όλοι όταν δισεκατομμύρια δολάρια από τις Ηνωμένες Πολιτείες διοχετεύονταν στην Αίγυπτο για υποστήριξη αυτού του καθεστώτος. Είμαστε υπέρ του λαού της Αιγύπτου που εξεγείρεται για τα δικαιώματα στην ευημερία, στην υγεία, στην εκπαίδευση. Γι' αυτό το λόγο πρέπει ομόθυμα το Κοινοβούλιο να συνεχίσει την στήριξή του θα πρέπει να πω ότι σε αυτή τη διαδικασία πρέπει να έχουμε έγνοια τους Παλαιστίνιους, να μην θυματοποιηθεί ο Παλαιστινιακός λαός. Εμείς, εκπροσωπώντας εδώ και την Κύπρο, μια γειτονική χώρα της Αιγύπτου, παρακολουθούμε τα γεγονότα με περισσή έγνοια και υποστηρίζουμε, επαναλαμβάνω, τα δικαιώματα του Αιγυπτιακού λαού σε αυτή την εξέγερση. Ευχαριστώ. E eh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Άστον, αγαπητοί συνάδελφοι, πραγματικά θα ήταν ευκταίο, όπω άκουσα και από άλλου, να μπορέσουμε να μπορεί να δημιουργηθεί ένα μέλλον δημοκρατικό για την Βόρεια Αφρική. Μια δημοκρατία όπω αυτή που έχουμε στην Ευρώπη. Όμω έχουμε και κινδύνου. Δεν μπορούμε αυτό να το, να το κρύβουμε. Όλοι θυμόμαστε την ε, απόπειρα που έγινε κατά των ε, κοπτών χριστιανών στην Αίγυπτο, ακριβώ τώρα, τα Χριστούγεννα. Θα πρέπει να καταφέρουμε να φτάσουμε. Τι συμβαίνει, δεν μακούτε; ακούτε, διακόπτη μιλήση. Μ' ακούτε, ωραία, ευχαριστώ. Λοιπόν, Συνεχίζω. Η φόβη μας είναι να μην, ε, να μην φτάσουμε σε μια Ισλαμική δικτατορία στη Βόρεια Αφρική. Και γι' αυτό η Ευρώπη θα πρέπει να είναι ο φύλακας να προσέξουμε να μην ε, επικρατήσουν Ισλαμικά καθεστώτα. Έχουμε ε, πολλέ πολλές εμπορικές σχέσεις με την Ευρώπη και αυτή, μέσα σε αυτή την οικονομική κρίση δεν θα είναι ευχάριστο να διακοπούν οι σχέσει αυτέ για την οικονομία μα και μην ξεχνάμε και τη μετανάστευση. Αυτή η αποσταθεροποίηση σίγουρα θα προκαλέσει αντίκτυπο κυρίω για τι χώρε στο νότο τη Ευρώπη. Και γι' αυτό ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την είπα το εκπρόσωπο να επαγρυπνεί για αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, Κυρία Άστον, να μην είστε τόσο αφελής, ούτε και εσείς κυρία Φέρχοφστατ, γιατί οι αδερφοί μουσουλμάνοι επιθυμούν το, τη Σαρία, που δεν είναι δημοκρατική. Ε, κυρία Άστον, ε, δεν άκουσα τίποτα σε σχέση με το Ισραήλ. Ε, μοιάζετε να είστε αφελείς και θέλετε ένα καλύτερο μέλλον για την Αίγυπτο, λέτε αλλά αρνείστε να αναφέρετε ρητά τον κίνδυνο που εκφράζει το Ισλάμ. Το Ισλάμ δεν είναι δημοκρατικό. Ε, κυρία Άστον, ε, δεν θέλουμε αφελείς πολιτικούς που πάνε στην Αίγυπτο με στρεβλά πολιτικά μηνύματα. Κυρία Άστον, να αντικρίσετε επιτέλους τον κίνδυνο που μας επαπειλεί. Και ε, παρακαλώ να προεδοποιήσετε τον Αιγυπτιακό λαό ότι ο Ισλαμικός νόμος είναι ένας τεράστιος κίνδυνος για όλους. Το ερώτημα το οποίο θα ήθελα να θέσω είναι, λέει ο κύριο Ντίβα, είναι το πώ μπορεί να ανθίσει η δημοκρατία σε κοινωνίε, όπου δεν υπάρχουν δημοκρατικοί θεσμοί και δεν υπάρχουν δημοκρατικές παραδόσεις. Η δημοκρατία δεν ξεπετάγεται ξαφνικά, δεν φυτρώνει σε ένα άνυδρο χωράφι. Πώς μπορεί λοιπόν να υπάρξει δημοκρατία εφόσον δεν υπάρχουν οι θεσμοί πάνω στους οποίους θα αναπτυχθεί. ο Δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω φυσικά με τον κύριο Ντίβα. Η δημοκρατία από τη μια μέρα στην άλλη δεν μπορεί να ξεπεταχτεί από το έδαφος. Χρειάζονται διαφορετικές προτεραιότητες στη συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν είμαι εγώ αυτός ο οποίος θα πει ποιος θα πρέπει να αναλάβει την Αίγυπτο. Οι Αιγύπτιοι θα πρέπει να επιλέξουν ανθρώπους οι οποίοι να μην είναι οι αδελφοί μουσουλμάνοι. Ο μαύρο; ένα μισή λεπτό. Βαρονιάστον. Δεν ήμουν πάντα πολύ ευγενής απέναντί σας. Πρέπει να αναγνωρίσω όμως ότι η ιστορία σας παίζει δύσκολα παιχνίδια και σας κάνει τη ζωή δύσκολη. Ελπίζω αυτά που ακούτε εδώ να μπορέσουν να σας βοηθήσουν. Το πρώτο πράγμα που θα ήθελα να υπογραμμίσω είναι ότι τα κράτη-μέλη δεν είναι αφέντες των πολιτών τους, αλλά εγγυητές της ζωής των πολιτών τους. Όταν από εγγυητές γίνονται αφέντες, τότε σταματάνε οι κυβερνήσεις και έρχονται τα καθεστώτα. Αυτό συνέβη στην Τινησία, αυτό συνέβη στην Αίγυπτο, πολιτικές ε, εμπειρίες οι οποίες συνόδευσαν ρομαντικά θα έλεγα την απελευθέρωση κράτησαν στις χώρες αυτές για δεκαετίες ολόκληρες και εμείς ε, υποστηρίξαμε τα καθεστώτα αυτά εις βάρος αυτών που διαδηλώνουν σήμερα. Δεύτερον, εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουμε μια ουσιαστική ευρωπαϊκή στρατηγική για την Μεσόγειο έχει αποτύχει δυστυχώς η διαδικασία για τις Βαρκελόνης και η Ένωση για τη Μεσόγειο. Είναι διακοσμητικά παιχνίδια αυτά. Δεν χρησιμεύουν σε κανέναν, δεν έχουν δημιουργήσει τίποτα και γι' αυτό θα πρέπει να τα καταγγείλουμε. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε από το μηδέν, θα πρέπει να σκεφτούμε μια νέα στρατηγική, να την κάνουμε πραγματικότητα, όπως το κάναμε και για την Ανατολική Ευρώπη, όπως το κάναμε έστω και με δυσκολίες για το συμφέρον των Βαλκανίων. Λοιπόν, δεν έχει σημασία το να λέμε θα μιλήσουμε με μία φωνή, γιατί τότε φοβάμαι ότι η φωνή αυτή δεν θα λέγει τίποτα. Παντσέρι δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Κύριε Άστον, έχω την εντύπωση ότι από πλευρά σας δεν υπάρχει μια συνειδητοποίηση ουσιαστικά του τι συμβαίνει στη Μεσόγειο. Νομίζω ότι μόνο αυτή η έλλειψη επαφής με τις εξελίξεις εξηγεί θα έλεγα τις ε, θέσεις που δεν έχουμε ουσιαστικά απέναντι στις αλλαγές. Έκλεισε η ιστορική φάση η οποία χαρακτήρισε μια Ευρώπη με μια πολιτική σύγχυση απέναντι στον Νότο και σε οικονομικό επίπεδο και στήριξης των ε, αρχών των χωρών αυτών και αντιμετώπισης ε, ε, άτακτης, θα έλεγα, του προβλήματος της μετανάστευσης. Νομίζω ότι δεν θα πετύχουμε τίποτα αν θεωρούμε ότι θα πρέπει να υποστηρίξουμε μόνο ε, απλά τις εκδηλώσεις, τις λαϊκές και τις διαδηλώσεις. Πρέπει να είμαστε ενήλικες πολιτικά, πρέπει να συντονιστούμε πολιτικά. Οι υπεύθυνοι για την εξωτερική πολιτική πρέπει να φύγουν ουσιαστικά από μια ημιπαρανομία μέσα στην οποία λειτουργούν και να συνοδεύσουν τις διαδικασίες που έχουν αρχίσει να εξελίσσονται. Απαιτείται μια νέα πολιτική γειτονίας, μια νέα πολιτική ασφάλειας με τη Μεσόγειο, μια διαφορετικού τύπου διαθεσιμότητα του συνόλου της Ευρώπης για την αντιμετώπιση του προβλήματος στη Μεσόγειο μια πολυ, αντιμετώπιση σε συνεργασία με την Τουρκία και με τις Ηνωμένε Πολιτείες. Είναι απαραίτητο να αλλάξουμε δρόμο στην πολιτική μας και γι' αυτό νομίζω ότι θα ήταν ιδιαίτερα τίμιο από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ξεκινήσει ένα νέο κεφάλαιο στην εξωτερική μας πολιτική απέναντι στη Μεσόγειο. Να τεθεί το θέμα της Ένωσης για τη Μεσόγειο αλλά ταυτόχρονα η Ευρώπη να είναι παρούσα στη Μεσόγειο. Αυτό είναι χρήσιμο για την Ευρώπη και δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Η κυρία δυόμιση λεπτά. Ο κόσμος αλλάζει. Ιδιαίτερα ο αραβικός κόσμος όπου το 40% του κόσμου ζει κάτω από το όριο της φτώχειας και το ποσοστό ανεργίας των νέων είναι το υψηλότερο στον κόσμο θέλουν την ανάπτυξη, θέλουν την δημοκρατία, αυτά πάνε μαζί. Και στην Τινησία και στην Αίγυπτο οι λαοί αυτοί αποφάσισαν να αναλάβουν οι ίδιοι τις τύχες τους για να προκαλέσουν τις αλλαγές που χρειάζονται. Οι κινήσεις αυτές, παρόλες τις προκλήσεις όπως είδαμε σήμερα στο Κάιρο και παρόλες τις δυσκολίες, τα κινήματα αυτά κανείς δεν θα μπορέσει να τα εμποδίσει. Για την Τινησία χθε και για την Αίγυπτο σήμερα υπάρχει μία φωνή την οποία ακούσαμε, είναι η ΙΠΑ οι ΙΠΑ υποστήριξαν ξεκάθαρα τους δημοκράτες. Εγώ πιστεύω στην Ευρώπη. Πιστεύω ότι έχει νόημα η Ευρώπη μόνο αν και αυτή αποφασιστικά στηρίζει πάντα και συστηματικά τους δημοκράτες. Θα ήθελα η Ευρώπη αυτή να είναι παρούσα στο ραντεβού με την ιστορία. Δεν ήτανε, δεν φταίτε μόνο εσείς. Αλλά φταίνε και οι φοβίες των ηγετών της Ευρώπης που προτιμούν την ακινησία και όχι την κίνηση. 20 χρόνια μετά από την πτώση του τείχους ζούμε μια νέα ιστορική αλλαγή. Συνειδητοποιήστε το. Αν δεν το κάνετε θα χάσετε και αυτό το ραντεβού με την ιστορία. Ευχαριστώ κύριε Σίπινγκ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κοιτάξτε, όλα αυτά που θέλω να πω ήδη υπόθηκαν. Απλώ μια ερώτηση λοιπόν θα θέσω στην ύπατη εκπρόσωπο. Σήμερα ο κύριο Μπλέρο, ο Τόνι Μπλέρο, πρώην πρωθυπουργό τη Βρετανία, τον οποίο πιθανότατα γνωρίζετε, είχε επενέσει επένεσε τον Χόσνι το το CNN το είπε. Είπε ότι ο Μπομπάραξ είναι πραγματικά ε, θαραλέος. Επίσης, ε, προειδοποίησε ότι πρέπει να γίνουν γρήγορα εκλογές στην Αίγυπτο. Τώρα ο κύριο Μπλερ είναι απεσταλμένο ε, για την ειρηνευτική διαδικασία Ισραήλ-Παλαιστίνη που στηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι είναι, ποια είναι η αποψή σα για τις δηλώσεις του Τόνι Μπλερ. Ο κύριος Μπάτον για ένα λεπτό. Η Αίγυπτος και για οι άλλες βορειοαφρικανικές χώρες δεν θα δουν ε, δυτικού τύπου δημοκρατίες ε, αλλά μάλλον ε, Ισλαμικό νόμο και νέο μεσαίωνα όπως είδαμε στο Ιράν. Ωστόσο υπάρχει μια ικανοποίηση που μπορεί κανείς να αντλήσει από τη διαδικασία καταπιεσμένων λαών που ανατρέπουν τα μη κυβερνητικά αυτά και πολιταρχικά καθεστώτα και μπορεί κανείς να καταπιέζει ένα λαό για τόσο καιρό και τόσο πολύ που πάντα να υπάρχει δυνατότητα να αντιδράσουν και να επαναστατήσουν. Υπάρχει τώρα εδώ μια αντίστοιχη ιστορία με τη Βρετανία όπου οι υποτυχείς κυβερνήσεις όλων των πολιτικών χρωμάτων πρόδωσαν τη χώρα μας και έδωσαν τα, τα δικαιώματά μας για αυτό διάθεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, οι Άγγλοι είχαν το δικαίωμα παλιότερα της ε, νόμιμη ε, επανάσταση. Δεν ξέρω πόσο μπορεί κανείς ε, να του στύψει ακόμα μέχρι να βγουν στους δρόμους όπως οι Αιγύπτιοι. Ο κύριος Μπρόνς, όλοι βέβαια χειροκροτάμε την ανατροπή καταπιεστικών καθεστώτων, αλλά μόνο όταν γνωρίζουμε ποιοι θα τους αντικαταστήσουν. Στην την Ισία, όπως και στην Αίγυπτο, ήταν καταπιεστικό το καθεστώς, ακόμα και με τα στάνταρ της Μέσης Ανατολής, αλλά και πάλι ήταν κοσμική, και σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση, υποτίθεται. Όμως ε, αυτό το πολιτερχικό καθεστώς μπορεί να αντικατασταθεί από κάτι πολύ χειρότερο. Μια πολιτισμένη μεταφορά εξουσίας σε όλες αυτές τις χώρες ε, ε, δεν νομίζω να υπάρχει. Δηλαδή όσοι μπορεί να το σκέφτονται, ας το ξανασκεφτούν. Επίσης θα πρέπει να σκεφτούμε ότι ε, οι οικονομίε των χωρών αυτών θα καταστραφούν και οι πληθυσμοί μας μπορεί να στείλουν βοήθεια, αλλά όχι να στείλουμε και στρατεύματα δικά μας εκεί να ε, ε, σκοτωθούν. Θα πρέπει να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους λαούς αυτών των χωρών. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ο κόσμος και η Ευρώπη όλος ιδιαίτερος δεν μπορούν να μείνουν αδιάφοροι απέναντι σε μια ε, λαϊκή επανάσταση που γίνεται στις χώρες της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής και κανείς δεν αμφισβητεί την νομιμότητα αυτών των διαδηλώσεων. Ένας λαός που διεκδικεί την ελευθερία του, μόνο αλληλεγγύη μπορεί να δει από εμά. Το ίδιο κάναμε και στο παρελθόν με τους φίλους μας της Ανατολικής Ευρώπης. Αυτή τη στιγμή ζούμε μια σπάνια στιγμή της ιστορίας και πρέπει να επιβεβαιώσουμε αντικειμενικά ότι ο εξτρεμιστικός Ισλαμισμός ε, θα πρέπει να δώσει πολιτική απάντηση και όχι θρησκευτική στα προβλήματα αυτά και να μην ε, οδηγήσει σε κοινωνικό απεκλεισμό. Θα πρέπει να γίνει μετάβαση προς ε, στέρεες δημοκρατίες που θα σέβονται τις μειονότητες είναι ένα μέρος του κόσμου που θα πρέπει να εκμεταλλευτεί αυτή την ε, φάση αναγέννησης για να προχωρήσει ειρηνικά στην ε, ευημερία. Ανεξάρτητα από την ε, θρησκεία του, τις πολιτικές του πεποίθησεις, όλοι, να μπορέσουν, όλοι εκεί να μπορέσουν να συγκατοικήσουν ειρηνικά. Και, και τελειώνω λέγοντας ότι θα πρέπει όλοι μαζί Ε, με μία φωνή λέμε στα πορτογαλικά ότι πρέπει να είναι πολύ δύσκολο να είναι κανείς ε, παπάς σε αυτή την ενορία αλλά θα πρέπει να προσπαθήσετε να μιλήσετε με μία φωνή χωρίς ριζοσπαστισμούς ε, και να υποστηρίξετε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σας ευχαριστώ. Αλκαντράου για δύο λεπτά. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Ήπατη εκπρόσωπη, αγαπητοί συνάδελφοι, αυτή τη στιγμή λαμβάνουν χώρα βίες αντιπαραθέσεις, βίες συγκρούσεις μεταξύ των υπαρασπιστών και των πολέμιων του Μουμπάρακ και νομίζω ότι θα πρέπει εμείς να δώσουμε ένα ξεκάθαρο σινιάλο προς τον ε, Μουμπάρακ και τους υποστηρικτές τους. Δηλαδή να αποχωρήσει άμεσα χωρίς να χυθεί παραπάνω αίμα. Αυτό το οποίο συνέβη στην Αίγυπτο μας κατέπληξε όλους, αυτό υπόθηκε ήδη. Αλλά θα πρέπει να το δούμε σαν μια ευκαιρία αυτή η περιοχή μετά από χρόνια πολιτικής και οικονομικής στασιμότητας να μεταβεί σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα. Ε, οι νέοι, ε, τα εκατομμύρια νέων επιθυμούν ε, να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε τις συνέπειες. Ορισμένοι κάνουν μια σύγκριση με το 89 ε, ένα 89 για τον ευρωπαϊκό κόσμο. Θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να υποστηρίξει στεναρά τον εκδημοκρατισμό. Θα πρέπει να καταστήσουμε άμεσα σαφές ότι αυτή η μεταβατική φάση θα πρέπει να ξεκινήσει άμεσα και ο Μουμπάρακ δεν έχει πλέον την νομιμότητα να ηγηθεί αυτή τη ε, διαδικασία εκδημοκρατισμού. Χρειαζόμαστε ή δυνατόν άμεσα ένα ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση μέτρων που θα έχουν σαν αποτέλεσμα την διενέργεια των πρώτων ελεύθερων και διαφανών εκλογών. Δηλαδή, μεταξύ άλλων, μια αλλαγή του συντάγματος, μια αλλαγή του εκλογικού δικαιώματος και μια αλλαγή της ε, αντιμετώπισης τάσης εναντί των ε, ΜΜΕ ούτως ώστε να μπορούν ε, να θέσουν υποψηφιότητα όσοι το επιθυμούν. Νομίζω ότι θα πρέπει οι δημοκρατικές δυνάμεις να υποστηριχθούν και η Ευρώπη καλύτερα να διαδραματίσει ένα θετικό ρόλο. Αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε την πολυπλοκότητα αυτής της κατάστασης. Οι ένοπλες δυνάμεις, για παράδειγμα, θα ε, επενείται για τον προστατευτικό της ρόλο. Αλλά ταυτόχρονα είναι και ένας οικονομικός, οικονομικά σημαντικός παράγων ε, και θα είναι, είναι αναγκαίο να γίνουν και οικονομικές ε, μεταρρυθμίσεις. Ευχαριστώ. Ναι, κυρία είπα ότι εκπρόσωπε, αξιότιμη. Εξότιμη κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ακούω προσεκτικά τα όσα υπόθηκαν από την ύπατη εκπρόσωπα και από τους συναδέλφους. Πολλοί λένε ότι πραγματικά ε, εντυπωσιάστηκαν από τα τεκτενόμενα, από τα συμβάντα στην Αίγυπτο και στην ε, Νησία. Και αυτό μου κάνει εντύπωση, γιατί κατ' ουσία γνωρίζαμε ότι δεν πρόκειται εκεί για δημοκρατικά καθεστώτα, αλλά αντίθετα ε, πρόκειται για πολιταρχικά καθεστώτα τα οποία καταπίεζαν τους λαούς τους. Ε, ε, δεν θελήσαμε να το δούμε, δεν κάναμε τίποτα για να αλλάξει η κατάσταση. Θεωρήσαμε ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος να έχουμε σταθερότητα με, το, με την περιοχή και το χώρο της Μεσογείου. Αλλά κατέστη σαφές ότι η υποστήριξη αυταρχικών και διεφθαρμένων καθεστώτων ε, στο όνομα της σταθερότητας και στο όνομα της αποφυγής του χάος ε, τελικά οδηγεί σε αστάθεια με περισσότερο χάος και χωρίς καμία δυνατότητα για το μέλλον. Και ελπίζω ότι θα δείξουμε αρκετή σύνεση, που ώστε να στηρίξουμε τη διαδικασία και δημοκρατισμού. Και ιδιαίτερω θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σα στην ε, στήριξη των διαφόρων πολιτικών κομμάτων τόσο στην Τινησία όσο και στην Αίγυπτο. Γιατί είναι αδύναμα ε, κόμματα τα οποία τα τελευταία χρόνια δεν είχαν τη δυνατότητα να οργανωθούν και συνεπώ χρειάζονται τη δική μα βοήθεια για να μπορέσουν να διαδραματίσουν ένα καθοριστικό ρόλο ε, στι εκλογέ που ελπίζω να λάβουν χώρα σύντομα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σε αυτή τη φάση της συζήτησης ένα σημείο θέλω να θέσω. Επανειλημμένα Είδαμε εμείς τα καταφύγια των χωρών μας στη Δύση να γίνονται αντικείμενοι κατάχρησης από ακραίους οι οποίοι επιστρέφουν στις χώρες τους. Ε, χθες ήταν θα έλεγα τα 32 χρόνια από τότε που επέστρεψε ο Αγιατολά Μεϊνή από το Παρίσι στην Τεχεράνη. Είδαμε που μας πήγε αυτό. Αυτός που θέλει να διαλυθεί επίσης το Ισραήλ, ο Γκανούση, ε, επέστρεψε στην Τινησία μετά από 20 χρόνια, υποστηρίζει το Χαμάς, ε, το οποίο είναι στην ουσία παρακλάδι των αδελφών μουσουλμάνων. Στην ουσία λοιπόν η Αίγυπτος είναι η βάση αυτών των οργανώσεων, οι οποίοι προσπαθούν μέσω της τρομοκρατίας να επικρατήσουν. Πρέπει λοιπόν να πάρουμε σοβαρά μέτρα έτσι ώστε να πάψει η εκόλαψη των τρομοκρατών στις ίδιες μας τις χώρες και να στηρίξουμε δημοκρατικές κοινωνίες σε χώρες όπως η Αίγυπτος και η Τινησία με σωστά στοχευμένη οικονομική βοήθεια. 1,5 λεπτό κύριος Μπονσινιόρα. Signor Συμφωνώ με αυτά τα οποία είπαν οι συνάδελφοι του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Θα πρέπει να υποστηρίξω όμω ότι τα τελευταία συμβάντα στη Μεσόγειο προκάλεσαν σε όλους μα τεράστια έκπληξη. Μέχρι πριν λίγες εβδομάδες δεν είχαν προβλεφθεί τέτοιου τύπου εξεγεύσεις. Η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης υπό τη Βαρόνη Άστον και αυτή φαίνεται ότι εξεπλάγει και αποδεικνύει μια πολύ ασθενέστατη θα έλεγα ικανότητα αντίδρασης. Διαρωτώ με αν αξίζει τον κόπο να ξοδεύουμε τόσα χρήματα για μια υπηρεσία οργανωμένη με τον τρόπο αυτό. Στην ουσία βλέπουμε ότι υπάρχει μια πλήρης απουσία ευρωπαϊκής διάστασης στην μεσογειακή σκακέρα. Εμείς είμαστε υπέρ της αυτοδιάθεσης των λαών μέσω ελεύθερων εκλογών και όχι μέσω ενεργειών που επιβάλλονται από βίαιους εξτρεμιστές. Είναι ανάγκη η σταθερότητα να συμβαδίσει με τη δημοκρατία. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν έστω και καθυστερημένα να βοηθήσουμε την ενίσχυση της δημοκρατίας, την ελεύθερη πολιτική, το κράτος δικαίου και την ασφάλεια των πολιτών όλος ο κόσμος και εμείς οι Ευρωπαίοι σήμερα έχουμε ανάγκη από μια Μισόγειο η οποία να είναι και να ζει σε ειρήνη, να είναι ειρηνική και να ζει σε ειρήνη. Και θα πρέπει να πάρουμε όλα τα μέτρα για να βοηθήσουμε με στοστό τρόπο τις ε, οικονομικά όλες τις χώρες της Μεσογείου. Mrs. Romero, for one Κυρίες και κύριοι, οι δημοκράτες της ε, Τινησίας μας έδωσαν ένα μάθημα οριμότητας και δημοκρατίας αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε τις σφαγές που γίνονται στην Αίγυπτο ε, και θα πρέπει να μιλήσουμε με μία φωνή στην ε, Ευρώπη για να μπορέσουμε να σταματήσουμε αυτές τις σφαγές και να υπάρξει δημοκρατική αλλαγή και στην Αίγυπτο. Αλλά στην Τινησία ε, ε, αντιδράσαμε έγκαιρα. Θα προετοιμάσουμε ένα ψήφισμα, ε, θα αποσταλεί μια αντιπροσωπεία στην χώρα και είναι σημαντική η στήριξη προς τη χώρα αυτή, πρώτα στην Τινησία και μετά στην Αίγυπτο και προς όλες τις χώρες που ζητούν την ελευθερία. Γιατί μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα, γιατί η οικονομική κατάρρευση θα πρέπει να έχει το μικρότερο δυνατό κόστος. Υπάρχουν ορισμένοι που επιθυμούν ένα διαφορετικό μοντέλο ε, για την Τινησία από εμά. Ζούμε το τέλος της ε, απεικιοκρατίας και την αρχή μιας νέας εποχής ανεξαρτησίας. Το παράδειγμα της Τινησίας ε, μας δίνει τη δυνατότητα να σκεφτούμε ότι οι θέσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας μπορούν να αλλάξουν. Ε, η κυρία Σάκε για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κυρία Υπατή εκπρόσωπε. Έτσι όπως βρισκόμαστε εδώ, πολίτες στην Αίγυπτο ε, δέχονται επιθέσεις στην ε, πλατεία Ταχρήρ και ο στρατός δεν τους προστατεύει αλλά τους επιτίθεται. Στη διαδικασία ειρήνευσης υπάρχουν διαφορετικά ένα διαφορετικό υπόβαθρο. Ε, δημοκρατική διακυβέρνηση, κοινωνιοοικονομική εξέλιξη, όλοι αυτοί είναι σημαντικοί παράγοντες. Κυρία Πρόεδρε, αυτή είναι η σκοπή του προγράμματος Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή αυτή 3 ε, δισεκατομμύρια ευρώ δαπανήθηκαν από την Κομισιόν ε, για το σκοπό αυτό τα τελευταία 15 χρόνια. Και επειδή τα αιτήματα των πολιτών ευθυγραμμίζονται με τους πολιτικούς μας στόχους, διερωτώμε γιατί είναι τόσο δύσκολο να ε, κάνουμε στεναρές δηλώσεις, γιατί η ανάγκη αυτή η ανάληψη ενεργητικής δράσης είναι επιτακτική. Ε, γιατί υπάρχουν κάποια σύννεφα τα οποία διαιρούν ε, την Ευρώπη και αποδυναμώνουν τη δυνατότητα να αναλάβουμε δράση. Ε, θα πρέπει να δράσουμε άμεσα υποστηρίζοντα το λαό. Είναι τα δικά τους δικαιώματα και η εξεπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διακυβεύονται εδώ. Υπάρχει μια... Ε, η κυβέρνηση της ε, την Ισίας έκανε λογοκρισία στα σύγχρονα μέσα για να καταστήλει τους, ναούς, ε, τους λαούς. Η Vodafone είχε μια πολύ ισχυρή παρουσία στην Αίγυπτο εμποδίζοντας πρόσβαση σε αυτά τα μέσα. Θα ήθελα να γίνει μια διερεύνηση του ρόλου αυτών των εταιριών οι οποίοι παρεμπόδισαν την ελεύθερη έκφραση ούτως ώστε να υπάρξει επιτέλους ένα σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών. Unia Europejska w relacjach e, z Tunezją, z Egiptem, moim zdaniem, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είπατε η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε διάφορα λάθη στο παρελθόν στη σχέση μας με την Τινησία όταν ήμασταν ήσυχοι το 2009 και όταν ο Μπεναλή κέρδισε τις δίθεν εκλογές ε, με 90% ποσοστό αυτές οι εκλογές ήταν ελεύθερες και δημοκρατικές παρομοίως στην Ισία, ο ποινικό κώδικας μεταρρυθμίστηκε υποτίθεται όμως δεν επιτρέπεται καμία δραστηριότητα κοιό ή υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και σήμερα αυτή η παθητική πολιτική ε, απέναντι στη Βόρεια Αφρική είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε πλέον να συνεχίσουμε. Πρέπει να είμαστε αποφασισμένοι να αποκατασταθεί η σταθερότητα στην περιοχή, διότι χωρίς εμάς θα είναι αυτό πάρα πολύ δύσκολο. Μόνο η δραστήριά μας ε, και αποφασισμένη θέση απέναντι στην κατάσταση στη <coughs> Βόρεια Αφρική μπορεί να βοηθήσει την αποκατάσταση του κράτους δικαίου ο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ελευθεροτυπία. Okay. Αγαπητοί συνάδελφοι, συζητάμε εδώ τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τινησία. Και παλιότερα πάνω σε αυτό το θέμα έλεγα ότι τα κοινωνικά κεκτημένα των Τινησίων θα έπρεπε να είχαν συνοδευτεί από πολιτικά κέρδη. Έχουν υπάρξει λοιπόν τελευταία κάποιες πολιτικές εξελίξεις. Η εξέγερση εκφράζει την επιθυμία για ελευθερία των Τινησίων το ίδιο ισχύει και για την Αίγυπτο, αν και τα πράγματα τρέχουν ακόμα στην Αίγυπτο και δεν ξέρουμε ακριβώς τι θα γίνει και ποιοι θα αναλάβουν την εξουσία αύριο στο όνομα της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Κάποιοι από μας φοβούνται βέβαια ότι αυτός ο άνεμος ελευθερίας δεν θα οδηγήσει στη διατήρηση του λαϊκού χαρακτήρα του κράτους, στη μετριοπάθεια και στην σταθερότητα θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι είναι πάρα πολύ πιθανό τις επόμενες εβδομάδες, τους επόμενους μήνες η περιοχή αυτή να μην έχει καθεστώτα τα οποία να είναι πολιτικά σταθερά και φιλελεύθερα και να μην εμπνέονται από τις ιδέες της ελευθερίας και της μετριοπάθειας. Πρέπει να προετοιμαστούμε και για αυτήν την πιθανότητα. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να ενθαρρύνω την ε, ε, κυρία Άστον να, να προσδιορίσει την εξωτερική πολιτική μας στα πλαίσια των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2005 για τη συνάντηση κορυφής της Βαρκελόνης. Ο κύριος Σαρίφ, δύο λεπτά. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, μέχρι τώρα πίστευα ότι οι λαοί είναι πρωτοπόροι σε σχέση με την πολιτική του ελίτ αλλά τώρα έχω και την απόδειξη. Να χαιρετήσω λοιπόν το θάρρος και την αποφασιστικότητα των Τινησίων και των Αιγυπτίων. Οι αξίες τις οποίες εμείς προσφέρουμε στον κόσμο είναι αξίες που δεν είναι μόνο δική μας όπως πιστεύουν ορισμένοι, αλλά είναι καθολικές αξίες τις οποίες όλοι συμμερίζονται. Η Ευρώπη δεν μπορεί νομίζω να συνεχίσει να συμπεριφέρεται σε αυτή την περιοχή του κόσμου με βάση λάθος αναλύσεις. Πρέπει να χαιρετήσουμε το, το θάρρος τους και τις προσδοκίες των λαών. Δεν είναι φιλανθρωπία, είναι ένδειξη ευθύνης. Σε αυτήν την αβέβαιη περίοδο κανένας δεν επιθυμεί το χάος και κανένας δεν επιθυμεί το status quo. Πρέπει εμείς να συνοδεύσουμε τα γεγονότα στην Αίγυπτο και στην Τινησία για να βοηθήσουμε τις δημοκρατίες που θα ωφελήσουν τις χώρες, τους πληθυσμούς τους και για μας τους ίδιους και νομίζω ότι το είπατε αυτό κυρία Άστον. Κλείνοντας θα ήθελα να επανέλθω σε αυτό που λέγανε ορισμένοι ότι οι λαοί μερικές φορές βρίσκονται σε στασιμότητα ακριβώς γιατί δεν βλέπουν στο μέλλον. Ελπίζω όμως ότι τώρα πια οι συνειδήσεις θα ξυπνήσουν. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κυρία Άστον. Θα ήθελα να σας πω να είστε πιο θαραλέα, να πάτε στο Κάιρο πριν από το Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών. Μιλήστε με του εκπροσώπου τη κυβέρνηση, με την αντιπολίτευση και όταν γυρίσετε στι Βρυξέλλε να μα εξηγήσετε τι ακούσατε. Να υλοποιήσετε την ε, ατζέντα. Ε, και ε, να μας δώσετε όλα τα στοιχεία ε, δεν είναι δυνατόν να αντιδρούν πρώτοι οι Αμερικανοί. Είστε η Ευρωπαία Υπουργό Εξωτερικών και θα ήθελα πραγματικά να συμβουλεύσω να το πράξετε άμεσα. Από την άλλη, ω Ευρωπαία Υπουργό Εξωτερικών, δεν θα πρέπει ε, να σας χορεύουν όλοι στο ταψί. Ε, θεωρώ ότι η πλατεία Ταχρίν το 11 είναι σαν την Αλεξάνδερ Πλάτς ε, του Βερολίνου το 89. Ε, εδώ έχουμε, λαμβάνει η χώρα μια επανάσταση. Εμείς θέλουμε δημοκρατία, ελευθερία και σταθερότητα και παραγνωρίζουμε ότι αυτή η διαδικασία μετάβασης από μια σταθερή δικτατορία προς μια δημοκρατία σπάνια γίνεται διαταγμένα, ειρηνικά και με σταθερό τρόπο. Και στο μέτρο αυτό και η διπλωματία και η οργάνωση αλλά και η προσοχή έχει τη θέση της. Ε, πρόκειται για μια επανάσταση κατά τη δικατορίας και υπέρ τη ελευθερία. Νομίζω ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να επιβάλλει τη δική τη βούλη σε αυτού του λαού. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Αλλά είναι ξεκάθαρο ότι μπορούμε να ασκήσουμε έστω περιορισμένα κάποια επιρροή. Δεν είναι δυνατόν να παραμείνει ο Μουμπάρακ, γιατί με την παρέμβαση του στρατού στην πλατεία Ταχρήρ έχει χαθεί και το τελευταίο κομμάτι νομιμότητα για τον Μουμπάρακ. Ο κύριος ε, Κάριμ. Αυτή η στιγμή την περιμέναμε από καιρό ε, και αυτοί ηγήθηκαν οι παλαιοί αλλά και αυτοί που δεν γνώρισαν τίποτα άλλο από το Μουμπάρακ στην Αίγυπτο. Η απάντησή μας ήταν να πούμε ότι η Αίγυπτος δεν θα έπρεπε να αποσταθεροποιηθεί περαιτέρω από ό,τι ήδη έχει αποσταθεροποιηθεί. Αλλά ο πληθυσμό τη ε, Αιγύπτου θα πρέπει να έχει την κυβέρνηση που επιθυμεί. Αυτό είναι ορθό, αλλά δεν επαρκεί και ε, σήμερα άκουσα φωνές προειδοποίησης ε, για τους Ισλαμιστές που ε, ελοχεύουν για να ορμήξουν και να πάρουν την εξουσία. δεν... Και δεν πρέπει να δώσετε καμία αξία στους, δεν δίνετε καμία αξία στους ανθρώπους που πλήρωσαν με τη ζωή τους στην Τινησία και στην Αίγυπτο το τίμημα της ανατροπής αυτών των καθεστώτων. Γιατί ε, εκείνοι στους δρόμους ε, εκτός του ότι είναι πολύ σε αριθμό είναι, η φωνή τους είναι ισχνή. Είπατε εκπρόσωπε ε, να έχετε ε, δύναμη στη φωνή σας να αποστείλετε ένα ξεκάθαρο μήνυμα γιατί ο Μουμπάρακ πρέπει να φύγει αμέσως. Ο κύριος ε, Μπούσατιλ. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η Ευρώπη θα πρέπει να κάνει πολλά περισσότερα για να δείξει στον αραβικό κόσμο το δρόμο για τη δημοκρατία. Όμως υπάρχει κάτι το θετικό που, που απορρέει από αυτά τα δραματικά γεγονότα, ότι οι λαοί ίδιοι που προέβησαν σε δράση θέλησαν να βελτιώσουν τη δική τους κατάσταση. Εξάλλου η ιστορία είναι γεμάτη από τέτοιες καταστάσεις και παρεμβάσεις ε, από τη Δύση που κατέληξαν να, να βλάψουν περισσότερο παρά να ωφελήσουν την κατάσταση. Αμείς, λοιπόν χρειάζεται... Παρέμβουμε για να γίνουν βελτιώσεις. Να γίνουν βελτιώσεις υπό το φως των γεγονότων που έχουν γίνει. Πρέπει να κάνουμε δύο πράγματα λοιπόν. Ε, καταρχήν να βοηθήσουμε εξίσου την πρόθεση της δημοκρατίας σε αυτές τις χώρες και όλος ιδιαίτερα στα δημοκρατικά ε, όργανα ώστε να μπορέσουν να ανθίσουν και να ανθίσουν με τέτοιο τρόπο ώστε οι εξτρεμιστές και οι νέοι δικτάτορες να μην μπορούν να βρουν πάτημα. Να διερωτηθούμε επίσης πού κάναμε λάθος. Μήπως η μεσογειακή μας πολιτική ήταν κενή περιεχομένου. Η Ευρώπη δεν μπορεί μόνο να αντιδρά, πρέπει να δράσει πια. Η Ευρώπη λοιπόν αυτή τη στιγμή προσπαθεί να στηρίξει τον ε, λαό της Τινησίας και τη μεταβατική κυβέρνηση στα πλαίσια του ευρωμεσογειακού διαλόγου που δεν πήγε καλά τα τελευταία χρόνια. Η έκρηξη οργής των νέων και των φτωχών του Μαγκρέπ και της Αιγύπτου προέρχεται από την άνηση κατανομή του πλούτου και από τον περιορισμό των δημοκρατικών ελευθεριών. Ο λαός ζητάει περισσότερη δημοκρατία, περισσότερη οικονομική ανάπτυξη, συμμετοχή στη δημοκρατία και εκπλήσεται όταν βλέπει την Ευρώπη, τη γυραιά Ήπειρο, ακίνητη, στάσιμη, ανίκανη να αναπτύξει ουσιαστικές πολιτικές ειρήνης. Η Ευρώπη στρέφει την προσοχή της βέβαια στην, στα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ζητά να υπάρξει πραγματικός διάλογος και πρέπει να ανοίξει ε, τα σύνορά της και να καταστήσει την Μεσόγειο μια θάλασσα ειρήνης και δεν θα πρέπει να συνεργάζεται με βίαιες χώρες στον τομέα των μεταναστών όπως η Λιβύη. Απαιτείται πιο ουσιαστική ευρωμεσογειακή πολιτική. Το απαιτεί η ιστορία. Το καλή η ιστορία. Σιωμπρό. Η κατάσταση στην Τινησία είναι κάπως διαφορετική βέβαια από αυτήν της Αιγύπτου. Οι αιτίε ίσως ε, να είναι οι ίδιες που οδήγησαν στις εξεγέρσεις στις δύο αυτές χώρες, αλλά οι συνέπειες στην εξωτερική πολιτική και στην ισορροπία της περιφέρειας θα είναι διαφορετικές. Πρέπει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί στην Αίγυπτο, για την Αίγυπτο. Ο Μουμπάρακ έδωσε κάποιες εγγυήσεις για την ασφάλεια της περιοχής. Η ανατροπή του σήμερα από ένα κίνημα το οποίο δεν έχει δημοκρατική βάση πίσω του θα μπορούσε να οφείσει την Αίγυπτο στα χέρια των αδελφών μουσουλμάνων. Συνεπώς πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί για τις συνέπειες αυτών των ε, εξελίξεων. Ξέρουμε ότι αν η Αίγυπτος συμμαχήσει με το Χαμά συνεχίσει να, διώχνει, να διώκει τους χριστιανούς αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το αποφύγουμε. Φυσικά αναγνωρίζουμε τα αρνητικά του καθεστώτος Μουμπάρακ, αλλά θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε και σωστές λύσεις στα σημερινά προβλήματα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Τόσα συμβαίνουν στην Αίγυπτο και στην Ισία είναι ιδιαίτερα σημαντικά και είναι δυνατόν αυτές οι διαδικασίες αλλαγής να επεκταθούν και σε άλλες ε, χώρες της ε, μεσογειακής περιοχής που είναι ιδιαίτερα σημαντική για την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί βρίσκεται στην άμεση γειτονία μας και έχουμε φιλικούς και στενούς δεσμούς με τις χώρες αυτές. Τα τελευταία δεκαετία Ευρωπαϊκή Ένωση Ένωση δεν μπόρεσε να πείσει τις αρχές της να προβούν στις ε, αναγκαίες μεταρρυθμίσεις. Στην ε, εσωτερική νομοθεσία, για παράδειγμα, εγώ επέμενα ότι η σταθερότητα δεν έπρεπε να χρησιμεύει σαν ε, άλοθη για μια στασιμότητα, αλλά οι χώρε αυτέ έπρεπε να κάνουν βαθιέ οικονομικέ και κοινωνικέ μεταρρυθμίσει. Τώρα τι μεταρρυθμίσει τι δουν οι πολίτε στο δρόμο. στο Συμβούλιο την ε, περασμένη Δευτέρα ε, ορίστηκε μία θέση ότι η διαδικασία μετάβασης ε, και θεωρούμε ότι η διαδικασία μετάβασης στην Τινησία πάει στη σωστή κατεύθυνση. αλλά τις τελευταίες εβδομάδες η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν απούσα. Ακούσαμε τις δηλώσεις του κ. Ομπάμα, ακούσαμε τις δηλώσεις της κ. Κλίντον. Επίσης εκπροσώπους του στρατού της Τινησίας οι νέοι μηχανισμοί της συνθήκης της Λισαβόνας θα έπρεπε να είναι πιο ορατοί. Κυρία Άστον, εγώ χαιρετίζω την επίσκεψή σα στην Τινησία σε δύο εβδομάδε, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να βελτιωθούν οι δυνατότητε πρόβλεψη και ταχεία αντίδραση. Θα πρέπει να διαδραματίσουμε ένα ενεργετικό ρόλο διεθνώ. Θα πρέπει να είμαστε σημαντικοί καταρχήν σε περιφερειακό και στη συνέχεια σε παγκόσμιο επίπεδο. Κυρία Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθεί του σύνεγγε στην κατάσταση στην Ισία και στηρίζει τι προσπάθειε του λαού για να υπάρξει μια ειρηνική μετάβαση προ τη δημοκρατία. Τα πρώτα μέτρα τα οποία υιοθετήθηκαν από τη μεταβατική κυβέρνηση πηγαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση και απευθύνουμε μια έκκληση προς τις αρχές ούτως ώστε οι αναληφθήσεις δεσμεύσεις πράγματι να υλοποιηθούν ούτως ώστε το κράτος δικαίου και οι θεμελιώδεις ελευθερίες πραγματικά να γίνουν σεβαστές και να υπάρξουν αληθινές πραγματικές μεταρρυθμίσεις σε οικονομικό και κοινωνικό πεδίο. Οι μεταρρυθμίσεις είναι το καλύτερο εργαλείο επένδυσης στο μέλλον και θα συμβάλλουν στην σταθερότητα και τη δημοκρατία σε αυτή τη χώρα. Η Ευρώπη επιθυμεί να έχει μια σταθερή εταιρική σχέση με την Τινησία στο πλαίσιο της Euromed και θα πρέπει να γίνουν ε, τα πάντα ώστε η διαδικασία μετάβαση στη χώρα αυτή να ενισχυθεί. Θα πρέπει ε, να δημιουργηθεί μια σταθερή δημοκρατία σε αυτή τη χώρα και θα πρέπει οι μεταρρυθμίσει να στηριχθούν από επαρκή οικονομικά μέσα. Θα πρέπει να ευημερήσει την Ισία, να είναι μια δημοκρατική χώρα και να μπορούμε να έχουμε μια καλή ε, συνεργασία που να δράσει στι κοινέ αξίε. Ο κύριο ε, Γκάλερ. Κυρία Πρόεδρε, εξότιμοι συνάδελφοι, αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε υπόθηκε κατ' επανάληψη. Εδώ υπάρχει πλουτιά συνένεση. Το ψήφισμά μα είναι ξεκάθαρο σε σχέση με την Τινησία. Για την Αίγυπτο θα πρέπει να γίνουν κάποιε προσθήκε με τι τροπολογίε. Νομίζω ότι υπάρχουν αρκετοί λόγοι για άσκηση αυτοκριτική. Η εκτελεστική εξουσία στι χώρε Μέλ και στι ε, έμειναν, ε, σε μια στάσιμη διατήρηση, ε, ε, σε μια στάσιμη κατάσταση και στο status quo θα έπρεπε να είχαμε απευθυνθεί νωρίτερα προς τις χώρες αυτές σχέση με τα δημοκρατικά ελλείμματα. Γνωρίζαμε ότι ε, ε, θα έπρεπε να έχει ασκηθεί αυτή η πολιτική, αλλά δεν είναι ακόμα πολύ αργά. Ο σεβασμός των ανθρωπίνων ε, δικαιωμάτων δεν σημαίνει παρέμβαση στα ιστορικά, στην ιστορική πολιτική των χωρών, αλλά ε, κανένα αυταρχικό καθεστώς δεν έχει εσωτερική σταθερότητα. Η Τινησία και η Αίγυπτος μπορούν να χρησιμεύσουν σαν παραδείγματα στις άλλες χώρες. Ορισμένοι φοβούνται να αναφέρουν ε, ονόματα άλλων χωρών. Για μένα, για παράδειγμα, η Σαουδική Αραβία θα μπορούσε να ακολουθήσει. Ωστόσο, οι 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν διαφορετικά συμφέροντα να μην, εάν έχετε τις ίδιες ε, ιδέες, παρακαλώ να αναλάβετε δράση. Αυτά, τα είπε, αυτά που είπε ο Ομπάμα χθε το βράδυ θα έπρεπε να τα είχατε πει εσείς. Θα πρέπει να χειραφετηθείτε εις όφελος Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτως ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να χαράξει τη δική της πολιτική γειτονίας. Ίσως την επόμενη εβδομάδα θα μπορούσατε να πάτε στην Αίγυπτο και στην Ισία και να μας πείτε την μεθεπόμενη εβδομάδα ε, να μας μιλήσετε σχετικά στην Ολομέλεια του Στρασβούργου ο κύριος Χάουιτ. Ε, θα πρέπει να εκδηλώσουμε την υποστήριξή μου μας στους ε, ειρηνικούς διαδηλωτές στην Αίγυπτο. Ε, επίσης θα πρέπει να μιλήσουμε για την Αλτζαζίρα. Συλλήφθηκαν έξι δημοσιογράφοι, ε, καθώς και για το θέμα του ίντερνετ, ε, της ε, της Vodafone από τη χώρα μου και άλλων εταιριών για τις επιλογές που έκαναν στην Αίγυπτο τις τελευταίες εβδομάδες. Επίσης ήθελα να πω ότι μα, Καλά θα ήταν οι Ευρωπαίοι ηγέτες να τα πούνε νωρίτερα αυτά που είναι σήμερα. Ο Σαρκοζή είπε το 2007 ότι θα ήθελα να πω, λέει, στον πρόεδρο Μουμπάρακ πω εκτιμώ την εμπειρία του, τη σοφία του. Ε, ο πρόεδρος Μουμπάρακ είναι φίλος μας. Ε, σήμερα ζητά την ε, αλλαγή. Ήθελε τη σταθερότητα, λέει, στην Αίγυπτο. Δεν είπε όμως πόσο θα ήθελε να γίνουν οι εκλογές και σήμερα πάλι ζητάει, εκλογε... Ε, ζητάει αλλαγή. Συμφωνώ με την υπατή ε, πρόσωπο. Η Ευρώπη είναι, σωστή, είναι καλή στην μεταβατική δικαιοσύνη, στην οικοδόμηση δημοκρατίας, στην ανάπτυξη της, κοινωνικής, ε, της κοινωνίας των πολιτών. Η Ευρώπη και εμείς θα πρέπει να δούμε μια, την κρίση στην περιοχή, αλλά σαν μια ευκαιρία για την Ευρώπη να αφιερώσει πόρου για να οικοδομήσει το σεβασμό για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτές ε, δεν είναι αρχές που επιβάλλουμε από την Ευρώπη. Αυτές τις ε, ζητούν στην Τίνιδα και το Κάιρο ο κόσμος που έχει κατεβεί στους δρόμους και είμαστε υποχρεωμένοι να το προσφέρουμε. Κύριο Σόνικ, 1,5 λεπτό. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κάθε επανάσταση ενέχει έναν κίνδυνο ότι η βούληση για δημοκρατία και ελευθερία θα ε, κλαπεί από από, τους, από άλλους. Ε, υπάρχει αυτός ο κίνδυνος στην Τινησία και στην Αίγυπτο, αλλά αυτό δεν πρέπει να, ποτέ ε, ε, ε, Λέσει λόγω να, να πάρουν την εξουσία οι Ισλαμικές δυνάμεις όπως έγινε στο Ιράν. Πραγματικά είναι μια δοκιμή για την Ευρώπη. Πρέπει να παίξουμε επιτέλους το ρόλο για τον οποίο υπάρχουμε. Να στηρίξουμε τις πολιτικές δυνάμεις που καλούν, που υποστηρίζουν την δημοκρατία και τον πλουραλισμό. Πρέπει επίσης να αναθεωρήσουμε την πολιτική γειτονία που μέχρι στιγμής εξυπηρέτησε αυτές τις διεφθαρμένες κυβερνήσεις. τα χρήματα που θα πρέπει να στηρίξουν την ευημερία του κόσμου εκεί θα πρέπει να κατευθυνθούν προς τις ΜΚΟ, τα πανεπιστήμια ε, και ούτω καθεξής. Θα πρέπει επίσης να στηρίξουμε προγράμματα για τους νέους και τις γυναίκες. Κυρία, είπατε εκπρόσωποι, η πολιτική μας αυτή τη στιγμή, σε αυτή την περιοχή του κόσμου, ε, μέχρι στιγμής δεν ήταν επιτυχία, ήταν αποτυχία. Θα πρέπει να διακινδυνεύσουμε, την, να υποστηρίξουμε την Αίγυπτο χωρίς το Μουμπάρακ σε δρόμο για μια κοσμική δημοκρατία της Αιγύπτου που θα σέβεται τις μειονότητες. Ο Μουμπάρακ πρέπει να φύγει. Είναι και η ώρα του. I Έχετε αγνοήσει, έχω ζητήσει το λόγο, λέει η κυρία Σίνκλερ. Η κυρία Σίνκλερ θέλει να θέσει μία ερώτηση. Παρακαλώ θα τη δεχτείτε. Κάνατε ορισμένα σχόλια δεν ξέρω αν ήσασταν νωρίτερα όταν κάποιος αναφέρθηκε στα σχόλια που έκανε ο κύριος Μπλερ. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με αυτά που είπε ο Τόνι Μπλερ. Χάουιτ. Λέω αυτά που είπα πάλι στην ομιλία μου. Νομίζω ότι από το παρελθόν πρέπει όλοι να βγάλουμε συμπεράσματα. Αλλά αυτό δεν πρέπει να μας σταματήσει σαν Ευρωπαϊκή Ένωση να ασχοληθούμε με την Αίγυπτο και τον αραβικό κόσμο στα πλαίσια της στήριξης της δημοκρατίας. Ελπίζω εσείς αν και έχετε διαφορετικές απόψεις για την Ευρώπη να συμφωνήσετε σε αυτό μαζί μου. Κυρία Βλάστο, πολλά ακούστηκαν Συμφωνώ πάντως με τις εκφράσεις συμπάθειας και εκτίμησης προς τους λαούς της Αιγύπτου και της Τινησίας, αντιπροσωπεύουν ένα σύμβολο ελπίδας για όλους. Θα ήθελα να πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία όπως είπαμε χαρακτηρίζεται από την απουσία της, πρέπει να βοηθήσει τους Αιγυπτίους και τους Αιγύπτιους για να μπορέσουν να ξεκινήσουν τις μεταρρυθμίσεις και να εγκαθιδρύσουν τη δημοκρατία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε ήδη να βοηθήσει τους Τινήσιους έτσι ώστε να προετοιμαστούν οι μελλοντικέ εκλογές, να κερδίσουν την δημοκρατία οι Τινήσιοι και να γνωρίσουν την κοινωνική ειρήνη και την ανάπτυξη με μια οικονομική ανάπτυξη που θα βοηθήσει τους νέους να δουλέψουν. Η, Ένωση... η Ένωση για τη Μεσόγειο ακριβώς νομίζω θα στηριχθεί και θα αναπτυχθεί από την Επανάσταση των λουλουδιών της Τινησίας. Η επανάσταση του Γιασεμιού λοιπόν θα οδηγήσει την Ευρώπη να βρει μια ισορροπία ανάμεσα στη μη επέμβαση στα εσωτερικά των χωρών αυτών αλλά και στη στήριξη της σταθερότητάς τους και της δημοκρατίας τους. Σβένσον. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εμείς ε, Μιλάμε συχνά για σεβασμό της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για ελευθερία. Και αληθεύει ότι συχνά Έχουμε ορίσει άλλες προτεραιότητες στο παρελθόν, όπως για παράδειγμα την πολιτική σταθερότητα. Τώρα, αναπάντεχα Βρισκόμαστε σε αυτή την κοινόπιν αυτή τη κατάσταση που και ο αραβικό κόσμο ζητά την ελευθερία και τη δημοκρατία και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Βεβαίω υπάρχουν κίνδυνοι έγινε λόγο ε, εντωμεταξύ για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των ελευθερίες που όλοι, ο, όλος ο κόσμος θα έπρεπε να χαίρει αυτών και τι θα γίνει τελικά. Θα πρέπει να τους ε, ε, διαβεβαιώσουμε ότι δεν θα κάτσουμε στην άκρη ως θεατές, αλλά ότι θα αναλάβουμε πρωτοβουλίες. Όπως είπε η Λέδη Άστον, πρέπει να είμαστε μέρος αυτής της οικοδόμησης της δημοκρατίας. Είναι εντυπωσιακό. Οι νέοι άνθρωποι ξεκίνησαν αυτή την επανάσταση και αυτό είναι κάτι που ίσως θα οφείλεται ε, στις δυνατότητες επικοινωνίας και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν πρέπει να τους επιβαρύνουμε με ιδεολογία και θρησκευτικέ ε, πεπιθήσεις. Μακρο, ε, τελικά στο κάτω-κάτω της γραφής η ελευθερία και τα ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει να επικρατήσουν και η δημοκρατία. Αυτό θα πρέπει να είναι το μήνυμα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Κυρία Ζαμπόρσκα, σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, κυρία είπατε εκπρόσωπε Λέδη Άστον, σας ευχαριστώ για χάρη μάλλον στην παρακολούθηση. Είδαμε στη, την υποβάθμιση της δημοκρατίας, την ε, έλλειψη ανεξιθρησίας στις χώρες τις οποίες συζητάμε και οι εκλογέ στις χώρες αυτές το αποδεικνύουν. Τα πολιτερχικά καθεστώτα δεν εμφανίζονται από μια μέρα στην άλλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κατάφερε να, να απαιτήσει ούτε καν την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δυστυχώ είμαστε οι τελευταίοι που φτάνουμε να και εκφράζουμε σε μια κοινή θέση. Και γιατί δημιουργήσαμε την Ευρωμεσογειακή Ένωση, δεν ε, είχαμε αρκετά διπλωματικά εργαλεία στη διάθεσή μα για να διαπραγματευτούμε την ειρήνη και τη σταθερότητα σε αυτό τι περιοχέ του κόσμου. Για δεκαετίε οι χώρε τη Ένωση στήριζαν αυτά τα καθεστώτα με οικονομικά μέσα κυρίω και τώρα οι ίδιοι σκέφτονται πώ θα παγώσουν τους, τη, την ε, βοήθεια και πώς θα υποστηρίξουν την αντιπολίτευση. Μα δεν είναι υποκρισία αυτό. Η κατάσταση στη Μεσόγειο είναι ένα δίδαγμα για μας για το μη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ελευθερία, ε, το, ανεξιθρησκεία δεν είναι σεβαστή. Μπορεί αυτό να αποτελέσει όπλο στα χέρια των ε, εξτρεμιστών. Και τα λέω όλα αυτά γιατί υπάρχουν και άλλες χώρες, πολλές ακόμη χώρες, που ακολουθούν το ίδιο δρόμο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Υπατή εκπρόσωπη, η συζήτηση εδώ σε αυτό το σώμα την ακολουθήσαμε με προσοχή και έχει κυρίως ένα κοινό παρανομαστή. Την, ε, το αίτημα προς εσάς, είπατε εκπρόσωπε, να υψώσετε τη φωνή σας, να προχωρήσετε προς τα μπρος, να είστε πιο θαραλέα να είστε πιο ηχηροί, να σταθείτε στο πλευρό ή να πάρετε το μέρος εκείνων που επιθυμούν μια σύγχρονη κοινωνία των πολιτών υπέρ της δημοκρατίας, της ελευθερίας της γνώμης και της ελευθερίας του τύπου. Η χώρα, η Τινησία και η Αίγυπτος βρίσκονται προ δύσκολων αλλαγών και χρειάζονται τη δική μας υποστήριξη. Δεν χρειάζονται αυτό που ακούω που άκουσε ο πρώτο σα εκπρόσωπο στη χώρα αυτή, ότι δεν χρειαζόμαστε καμία αλλαγή τη στρατηγική. Αντιθέτω, η στρατηγική για τη Μεσόγειο, ίσω η στρατηγική για την Εγγύη Ανατολή, ίσω η αναθεώρηση τη συνύπαρξη πέρα από τη Μεσόγειο και ε, πάντων η προετοιμασία των εκλογών και η υποστήριξη των εκλογών ε, θα πρέπει να έχει διαφύγει το εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χώρα αυτή ότι στην Ισία η μεταβατική κυβέρνηση θέλει να κάνει τέσσερις συμφωνίες για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την απελευθέρωση των, των πολιτικών κρατουμένων, την επιστροφή των αντιπολιτευόμενων, την διενέργεια ελεύθερων εκλογών. Αυτή είναι η διαδικασία που θα πρέπει να στηρίξουμε και το Κοινοβούλιο επιθυμεί από εσά μια πιο δυνατή φωνή. Ευχαριστώ κυρία Σκούρια για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κυρία ε, βαρώνει. Εμείς θέλουμε να καταλάβουμε γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν παίζει ένα πιο σοβαρό ρόλο στην εξωτερική πολιτική. Η εξωτερική πολιτική είναι κάτι το σοβαρό. Προβλέπει στρατηγικές, συγκεκριμένους στόχους και ξεκάθαρες συμμαχίες. Δεν μπορούμε να συνεχίζουμε να γυρνάμε στον κόσμο και να χτυπάμε την πλάτη ολονών φιλικά ε, ε, παριστάνοντας ότι όλα πάνε καλά. Δεν καταλάβαμε ότι αυτή η δικτατορία μας κοροϊδεύε όλους. Τώρα με χιλιάδες κόσμο στους δρόμους μιλάμε για δημοκρατία και για ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, εντάξει, ας έρθουν, αλλά ας βοηθήσουμε και να έρθουν, αλλά προσοχή. Προσοχή να μην ακολουθήσουμε τα πλήθη. Θυμάστε τον Ιρανικό λαό πώς ε, έδιωξε τον Σάχη και είδαμε πώς κατέληξε, πού κατέληξε η κατάσταση. Εγώ εύχομαι η νέα Αιγυπτιακή κυβέρνηση να μπορέσει να κρατήσει μακριά τους εξτρεμιστές, να παίξει το ρόλο που πρέπει στην Ισραηλοπαλαιστινιακή κρίση. Δημοκρατία περισσότερη, ναι, σε αυτό το μέρος του κόσμου, αλλά και περισσότερη ευρωπαϊκή πολιτική. Περνάμε στο Catch the Eye τώρα, όπως μπορείτε να φανταστείτε. Λάβαμε πάρα πολλά αιτήματα, δεν μπορώ να τα δεχτώ όλα. Ζητώ από όλους όσους ε, δώσω το λόγο να μείνουν στο λεπτό τους, στο ένα λεπτό τους, για να μπορέσουμε να ακούσουμε όσους γίνεται περισσότερο. Γιατί το πιο σημαντικό είναι βέβαια να ακούσουμε και την απάντηση της είπα της εκπροσώπου. Νικολάσιτς πρώτα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κυρία Υπατή, πρόσωπε υπάρχει μεγάλη ένταση στην Ισία και στην Αίγυπτο και αυτό ήταν αναμενόμενο ή θα έπρεπε να είναι αναμενόμενο γιατί τα προβλήματα στην οικονομία και στην κοινωνία είχαν αγνοηθεί για πολύ καιρό από τους κυβερνώντες. Συνεπώς είναι πολύ θλιβερό ότι υπάρχουν αυτές τις συγκρούσεις αυτή τη στιγμή αλλά αυτό υπογραμμίζει τη στιγμή, την ανάγκη να υποστηριχθεί η δημοκρατία απ' έξω ή τουλάχιστον δημοκρατικές δυνάμεις και αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι όλα τα υπάρχοντα εργαλεία για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το, το δικαίωμα της θρησκευτική ελευθερίας. Και θα πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι δεν θα ανεχθούμε ε, τους ε, αδιάλακτους Ισλαμιστέ να ανέλθουν στην εξουσία. Θα πρέπει να υποστηρίξουμε την κοινωνία των πολιτών, να υποστηρίξουμε τις αντιπολιτευτικέ δυνάμεις και την διενέργεια δημοκρατικών εκλογών. Το ότι συζητάμε το θέμα της Τινησίας όταν το θέμα της Αιγύπτου βρίσκεται σε σημείο βρασμού δείχνει πόσο καθυστερημένα αντιμετωπίζουμε την πραγματικότητα αν και ο τίτλος της συζήτησής μας αλλάζει εύκολα. Οι δημόσιες αντιδράσεις μας ήταν πάρα πολύ δειλές θα έλεγα. Στην ουσία εδώ γίνονται επαναστάσεις και εμείς συζητάμε να υπάρξει διάλογος. Οι προσδοκίες ότι οι επαναστάσεις αυτές θα οδηγήσουν σε δικές μας ε, ή μάλλον σε καταστάσεις που να εδράζονται με τη σειρά τους σε δικές μας αξίες θα διαψευστούν. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα σαν μια πρόκληση η οποία μας αναγκάζει να σταθούμε συντονισμένα και επικοδομητικά και όχι να λέμε μόνο καλά και ωραία λόγια. Εσείς θα πρέπει να υποστηριχθείτε κυρία Άστον από το Συμβούλιο στο σύνολό του χωρίς εξαιρέσεις. Θα πρέπει επίσης να ανησυχήσουμε για τα καθεστώτα τα οποία θα γεννήσουν οι καταστάσεις αυτές αφήνοντας βέβαια τους λαούς των χωρών αυτών να αποφασίσουν μόνοι τους. Στο Κάιρο ο λαός αποφάσισε ότι οι ηγέτες του και το πολιτικό του σύστημα δεν του αρκεί. Πολλοί υποστηρίζουν ότι ο Μουμπάρακ έπαιξε ένα πάρα πολύ θετικό ρόλο στη Μέση Ανατολή και υποτίθεται ότι βοήθησε στην σταθερότητα της περιοχής. Δεν με ενδιαφέρει αυτό όμως σε αυτή τη φάση. Τα γεγονότα της Τινησίας και της Αιγύπτου αποδεικνύουν την ανυπαρξία του ρόλου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συγγνώμη. Πρέπει να είναι πιο παρεμβατική η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθώντας να λυθούν τα προβλήματα στις περιοχές που μας περιβάλλουν όχι μόνο στο νότο της Ευρώπης αλλά και στην Λευκορωσία και στον Αγκόρνο Καραμπάχ. Νομίζω ότι θα πρέπει να κατανοήσουμε τον άνεμο της δημοκρατίας ο οποίος πνέει. Λέει Άστον πρέπει να φανείτε πιο φιλόδοξη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Άστον, Αφού κάναμε το σφάλμα να υποστηρίζουμε τα δικτατορικά καθεστώτα της Νοτιού Μεσογείου με το πρόσχημα ότι αποτελούν έναν άχωμα κατά του Ισλαμισμού. Σήμερα θα πρέπει να τεθούμε στο ύψος των ιστορικών στιγμών που διανύουμε. Η Ευρώπη θα πρέπει να χαράξει μια απαιτητική πολιτική εναντί των τυραννικών και δικτατορικών καθεστώτων. Ο Μουμπάρακ θα πρέπει να φύγει τώρα. Θα πρέπει να υποστηρίξουμε τη διαδικασία δημοκρατισμού που επέλεξαν οι λαοί. Θα πρέπει να είμαστε ε, σεμνοί. Οι διαδικασίες έχουν ξεκινήσει ήδη σε αυτές τις χώρες. Με συγχωρείτε λέει η ομιλήτρια. η οικονομική υποστήριξη θα πρέπει να επαναπροσανατολιστεί υπέρ των δημοκρατικών δυνάμεων. Ο κύριος, η κυρία Ματίας. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ πιστεύω πω αυτέ οι δύο χώρε, όπω και άλλε στην περιοχή, μα αποδεικνύουν ότι τα τελευταία χρόνια οι Ευρωπαίοι ηγέτε ε, τελικά ε, υποστήριξαν περισσότερο τι εμπορικέ συναλλαγέ και όχι τη δημοκρατία, υπέρ δηλαδή των ηγετών και, κατά, και όχι τόσο υπέρ των λαών. Πραγματικά ανησυχώ με τι εξελίξει στην Αίγυπτο, τι σημερινέ μάλιστα εξελίξει και όχι δεν πρέπει να είμαστε ηρεμοί, αλλά αλληλέγγυοι, αλληλέγγυοι με τα εκατομμύρια πολίτες ε, ε, Αιγυπτίων που έχουν κατέβει στους δρόμους στο Κάιρο σε ολόκληρη την ε, Αίγυπτο που έχουν κουραστεί από την καταπίεση και από την ανεργία και από τη φτώχεια ο Μουμπάρακ αφού έφτιαξε ένα καθεστώς και έφτιαξε έναν καθαρό και ανοιχτό δρόμο για την βία εμείς πρέπει να πούμε ότι πρέπει να σταθούμε στο πλευρό αυτών των ανθρώπων δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να επικρατήσει μια στατικική φόβους για να γυρίσουν σπίτι τους αν είχε γίνει αυτό στην Πορτογαλία θα είχαμε μείνει και εμείς σπίτια μας και ευτυχώς που δεν το κάναμε τότε γιατί ακόμα θα ήμασταν ε, γιατί σήμερα μάλλον έχουμε δημοκρατικό πια καθεστώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε που μου δώσετε το λόγο. Κυρία Άστον, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία διαθέτει πάρα πολλούς εμπειρογνώμονες οι οποίοι θα έπρεπε να είναι σε θέση να κάνουν μια επαγγελματική αξιολόγηση της κατάστασης για παράδειγμα στην Αίγυπτο και θα έπρεπε να είναι σε θέση να απευθύνουν κάποιες συστάσεις σε εσά εν σχέση με τα δυνατά βήματα τους ώστε να βοηθηθούν οι χώρες αυτές να απαλλαγούν από τους μη επιθυμητούς πολιτικούς ηγέτες η πολιτική στρουθοκομαλισμού ε, που πρεσβεύουμε ε, ε, μας κάνει να αμφιβάλλουμε κατά πόσο η υπηρεσία εξωτερικής δράσης είναι τόσο ικανή όσο θα θέλαμε. Κυρία Ήπατη, εκπρόσωπε της Ευρωπαϊκής Εάν διστάσουμε να δώσουμε μια στεναρή απάντηση στην κατάσταση στην Ισία και στην Αίγυπτο, οι φορολογούμενοι θα διαρωτηθούν γιατί πληρώνουμε όλους αυτούς τους ειδικού στην υπηρεσία εξωτερική δράση Ευρωπαϊκή Ένωση, αν δεν είναι σε θέση να παράσχουν επαγγελματικέ συμβουλές. Uh, Κυρία Άστον, οι αισιόδοξοι θεωρούν ότι τα επαναστατικά γεγονότα στην Αίγυπτο ή στην Τινησία προμηνύουν μια αραβική άνοιξη όπως ζήσαμε στο παρελθόν στην Ανατολική Ευρώπη. Εμείς ως Ευρωπαίοι στο, θα έπρεπε να είμαστε στο πλευρό της ελευθερίας και της δημοκρατίας και θα έπρεπε να, να χαιρόμαστε αν συνέβαινε κάτι τέτοιο. Αλλά θα πρέπει να λησμονούμε ότι εμείς οι Ευρωπαίοι της Δύσης ε, τελικά στηρίξαμε τους ε, αξιοθρύνητους αυτούς δικτάτορες. Δεν θα πρέπει να έχουμε ψευδεστήσεις. Το ίντερνετ και το Twitter είναι σύγχρονα μέσα για να προωθήσουν μια σύγχρονη επανάσταση αλλά δεν μπορούν να αντικαταστήσουν το κράτος δικαίου και και τις δημοκρατικές δομές που θα πρέπει να υπάρχουν πίσω από τα πρέπει να στα παρασκήνια για να στηρίξουν ένα δημοκρατικό καθεστώς, ε, τις δημοκρατικές δυνάμεις. Εμείς θα πρέπει να πάρουμε θέση και να εισφέρουμε στη δημιουργία τέτοιων δημοκρατικών δομών για την εμπέδωση του κράτους δικαίου και της ελευθερίας σε αυτές τις χώρες. Σας ευχαριστούμε η τελευταία, αυτή ήταν η τελευταία παρέμβαση του, στο πλαίσιο του Catch the Eye και τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Άστον για να απαντήσει. Σας ευχαριστώ πολύ. Να σας ξεκινήσω Καθιστώντα απόλυτα σαφές ότι δεν δέχομαι ότι η Ευρώπη ήταν αργή ή καθυστέρησε. Κάναμε αμέσω δηλώσεις και για την Τινησία στις 10 Ιανουαρίου. Εγώ έκανα δήλωση για την Αίγυπτο την περασμένη εβδομάδα πριν από όλου. Μα δεν είναι διαγωνισμός ούτε αγώνας. Αλλά δεν δέχομαι αυτή την επίκριση. Ούτε δέχομαι ότι αργήσαμε να ενεργήσουμε. Ήμασταν σε μόνιμη επαφή με την Τινησία και την Αίγυπτο με αποστολέ γραμμές μας εκεί και τις οποίες πρέπει και να τιμήσουμε ιδιαίτερα για τα όσα χρειάστηκε να κάνουν τις τελευταίες εβδομάδες και με τις υπηρεσίες μας ήμασταν σε διαρκή επαφή. Επίσης θα γνωρίζετε ότι είχαμε και άλλα θέματα με τα οποία ασχολούμαστε ταυτόχρονα. Δεν δέχομαι λοιπόν ότι ήμασταν πολύ ποιοι και ότι δεν, κάναμε, δεν ενεργήσαμε γρήγορα. Δέχομαι ότι πρέπει να κάνουμε και άλλα. Εσείς μου δώσατε όλα όμως τα εργαλεία που χρειάζομαι με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Πιθανότατα όχι. Τους πόρους που χρειάζομαι ούτε. Αλλά θα κάνουμε ό,τι μπορούμε μέσα στο πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί η εξωτερική υπηρεσία δράση και του ρόλου που έχω. Εγώ δεν είμαι κάποιο που μπορεί να βγαίνει και να λέει τι προσωπικέ του απόψει. Μιλώ εξ ονόματο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Σα ακούω εσά, ακούω τα κρατημέλη, ακούω και την Κομισιόν. Αυτό είναι ο ρόλο που εσεί σχεδιάσατε μέσα στη συνθήκη τη Λισαβόνα και αυτό και θα κάνω. Διότι όταν μιλώ με τον Τινήσιο Πρωθυπουργό και κάποιοι από εσά που δεν ήσασταν εδώ νωρίτερα, ήταν στο γραφείο μου σήμερα και έκανε την πρώτη του επίσκεψη εκτός ε, την Ισία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί εγώ τον κάλεσα και γιατί γνωρίζει πόσο σημαντικοί είμαστε εμείς, όχι μόνο σήμερα αλλά και αύριο μεθαύριο και τα επόμενα χρόνια. Και γιατί όταν του μιλάω εγώ είναι σαν να μιλάει ολόκληρη η Ευρώπη και γνωρίζει πολύ καλά ότι αυτά που εγώ λέω θα στηριχτούν από 27 χώρε και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από την Κομισιόν. Και αυτό σημαίνει κάτι για αυτούς τους ανθρώπους. Σημαίνει ότι όταν μιλάμε είναι ένα μήνυμα, όχι απαραίτητο όπως είπατε εδώ μια φωνή. Είναι όμως το ίδιο μήνυμα. Είτε το λέει ο καγκελάριος της Γερμανίας, είτε το λέει ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας, είτε ο πρόεδρος κάποιες άλλες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οποιοδήποτε από τους 27 ε, αντιπροσωπεύει όλους. Και γι' αυτό και οι Υπουργοί Εξωτερικών συγκεντρώθηκαν τη Δευτέρα και μετά από τα συμπεράσματα και τις, τα ανακοινοθέντα τύπου που έδωσαν για τη γειτονιά μας αλλά και πέρα από αυτή είναι τόσο σημαντικά για τον κόσμο επιτόπου. Και δεν θα πρέπει αυτό να το ξεχνάμε σε ό,τι κάνουμε. Συμφωνώ μαζί σα ότι πρέπει να είμαστε πιο δραστήριοι επιτόπου, να κάνουμε περισσότερα και συμφωνώ απολύτω ότι πρέπει να ξαναδούμε και να επανεξετάσουμε την πολιτική γυτνίασης. Το λέω εδώ και καιρό. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα είναι πιο διαφοροποιημένη η προσέγγιση μα, ότι κάθε χώρα θα την παίρνουμε και θα την βλέπουμε χωριστά και θα βλέπουμε τι θέλουμε να επιτύχουμε με το λαό τη τάδε και τη δύνας χώρα. Ναι, περισσότερα με την κοινωνία των πολιτών, ναι, περισσότερη έμφαση στα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία και να ε, ε, κοινά ζητήματα εξωτερική πολιτική συμφωνώ μαζί σα και προσπαθώ να το κάνω και αν δείτε τι κάνουμε του τελευταιου δυο τρει μήνε, θα δείτε κάτι το κοινό αυτά που λέω εγώ είναι περισσότερη δράση στην γειτονιά μα πρώτη προτεραιότητα μετά από την ε, δημιουργία τη Υπηρεσία. καλύτερη, ευφιέστερη και πιο σχετική πολιτική με τις ανάγκες τους Αξιότιμοι κύριε βουλευτέ, εγώ δεν μπορώ να αναλάβω την ευθύνη τώρα για το τι συνέβη πριν από τη δική μου ε, θητεία, αλλά αναλαμβάνω την ευθύνη να, να μετατρέψω αυτό το οποίο κληρονόμησα σε μια ευρωπαϊκή πολιτική. Και αυτό ξεκινά με τα όσα κάνουμε τώρα και πόσα θα μπορέσουμε να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και να προχωρήσουμε. Δεν υποτιμώ το πόσο δύσκολο, ε, δύσκολη και πόσο γρήγορη ε, με γρήγορα μεταβαλλόμενη είναι η κατάσταση. Συμφωνώ επίσης με εκείνου που τόνισαν πως η δημοκρατία δεν είναι μία στιγμή χρονική, είναι μία διαδικασία. Η δημοκρασία οικοδομείται βλέπεις ποιοι είναι οι οργανισμοί που μπορούν να συνεργαστούν με τον λαό, που, να κατα... που καταλαβαίνουν τα δημοκρατικά δικαιώματα, τι μπορούν να κάνουν με τα μόρφωση μιας ε, κοινωνίας. Τα χρησιμοποίησαμε αυτή τη λέξη αυτή τη λέξη στα συμπεράσματα του Συμβουλίου γιατί εγώ πραγματικά πιστεύω σε μεταμόρφωση και όχι αύριο αλλά μακροπρόθεσμα και αυτό προσφέρει η Ευρώπη. Προσφέρει και το προσέφερε και στα ίδια τα μέλη της. Έφερε την μεταμόρφωση που θα διαρκέσει για γενιές και γενιές. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Δεν θέλουμε να αντιδράσουμε άμεσα. Θέλουμε να δίνουμε κάτι το οποίο θα διαρκεί όχι για μία μονογενεά αλλά για πολλές περισσότερες. Και φυσικά δεν ξέχασα και όλα τα άλλα ζητήματα. Παρακολουθώ τι συμβαίνει. Ε, Φυσικά και ξέρω τι συμβαίνει στο Ιράν και την περασμένη εβδομάδα και την προπερασμένη ε, είχα συνομιλήσει με τους Ιρανούς και ξέρετε πόσο πολύ ε, με απασχολούν τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Ιράν λόγω των δηλώσεων που έχω κάνει και λόγω όλων των ε, ε, όσων συμβαίνουν εκεί. Για τη Μέση Ανατολή επίσης δεν το έχω ξεχάσει. Με τον Πρωθυπουργό θα μιλήσουμε αύριο. <coughs> Σίγουρα δεν το έχουμε ξεχάσει. Και εγώ θα προεδρεύσω του κουαρτέτου για την ασφάλεια στην Μέση Ανατολή. Ούτε την Αλβανία την ξέχασα. Ο Μύρος Λαφλάιτσεκ ήταν εκεί ε, αυτή τη εβδομάδα εκ, εκ μέρου μου για να ασχοληθεί με το θέμα. Κανένα από τα θέματα που συζητώνται εδώ στο Κοινοβούλιο απόψε. Και δεν είμαι υπεύθυνη φυσικά για τα τι είπε ο Τόνι Μπλερ. Μπορεί να μιλάμε την ίδια γλώσσα, να προερχόμαστε από το ίδιο πολιτικό κόμμα, αλλά δεν είμαι υπεύθυνη για αυτόν. Την επόμενη εβδομάδα θα πάω στο Συμβούλιο Ασφαλείας εξ ονόματος σας πάλι για να δείξουμε τι έχει να προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτούς τους λαούς για σήμερα και για αύριο. Και είναι πραγματικά πολύ σημαντικό να έχω την υποστήριξή σας για να το κάνω αυτό. Όχι, ησύχω μπορώ να είμαι και πολύ πιο ε, κραυγαλαία, ε, με, αλλά με συνοχή, με στόχους, με στρατηγική και σχέδιο. Έτσι ώστε όταν θα έρθει ο Αιγύπτιος Πρωθυπουργό στην γραφείο μου, να του δώσω και ένα σχέδιο. Δεν του πω καλώ ήρθατε, τι ωραία που σας, που σας βλέπω, ελάτε να μιλήσουμε πέντε λεφτά μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες. Όχι, ελάτε, καθίστε εδώ να δουλέψουμε το σχέδιό σας με το τι μπορούμε εμείς να προσφέρουμε, πόσα χρήματα, τι μπορούμε να κάνουμε, ποια μέσα χρειάζεται να συγκεντρώσουμε, πόση ευελιξία έχω στη διάθεσή μου, πόσα χρειάζομαι ακόμα, τι χρειάζεστε εσείς από εμά, από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, την, την Τράπεζα της Αφρικανικής Ένωσης, τη ΣΥΠΑ, πώς θα φτιάξουμε ένα πρόγραμμα και μετά ε, τον Πρωθυπουργό της ΕΜΕΝΣ να κάνουμε τα ίδια πάλι για να φτιάξουμε ένα νέο πρόγραμμα, ταμείο μάλλον αναπτυξιακό. Έτσι, κατά την άποψή μου, θα πρέπει να δουλεύει η Ευρώπη. Και αυτό κάνω καθημερινά εξ ονόματός σας και θα συνεχίσω και να το κάνω. Ελπίζω ότι θα μπορέσω να επανέλθω και να το συζητήσουμε εκ νέου αυτό το θέμα. Τα γεγονότα στην Αίγυπτο όμως εξελίσσονται με ταχύτητα και την ώρα που μιλάμε εμείς. Εμείς στείλαμε μηνύματα και προς τον Αντιπρόεδρο της ναι. Κυβέρνησης θα πρέπει οι δυνάμεις ασφαλείας ναι. φυσικά να σταματήσουν να ασκούν βία. Το μήνυμα το έστειλα ξεκάθαρα. Η κυβέρνηση είναι υπόλογη έτσι ώστε ο στρατός να βοηθήσει τους πολίτες και το λαό και να προστατεύονται οι πολίτες. Τα νοσοκομιακά θα, μπορούν να, θα πρέπει να μπορούν να φτάνουν στην πλατεία Ταχρήρ θα ξαναμιλήσω με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης μόλις φύγω από την αίθουσα. Υπάρχει μια συνάντηση η οποία προσπαθεί να βρει μια άκρη με τα κινήματα της αντιμοπολίτευσης. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες προσπαθούν να συνεργαστούν με άλλες ηγέτες του κόσμου έτσι ώστε να βρεθεί μια άκρη. Υπάρχουν διασταυρούμενες τηλεφωνικές κλήσεις ανάμεσα σε ηγέτες όπως ποτέ στο παρελθόν που καταλήγουν στην Αίγυπτο και ταυτόχρονα στα γραφεία μου υπάρχει μια συνεδρίαση η οποία ασχολείται με την κρίση στην χώρα αυτή. Αυτά κάνω λοιπόν καθημερινά εδώ από τότε που ξεκίνησε η χώρα αυτή και ταυτόχρονα με προβλήματα αντίστοιχα άλλη κλίμακας βέβαια στη Λευκορωσία, στην Αλβανία, στο Σουδάν και τα λοιπά. Αυτά κάνουμε. Αν μπορούμε να κάνουμε περισσότερα φυσικά. Προφανώς θα πρέπει να αποδώσουμε καλύτερα. Έχουμε κάνει όμως βήματα προόδου χωρίς να είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι. Το να φαίνομαι δεξιά-αριστερά ότι είμαι μαζί με όλους όσους θέλουν να φαίνονται δεν είναι αυτή η δουλειά μου. Εγώ θα προσπαθήσω να βοηθήσω αυτό το οποίο η Ευρώπη θέλει να πετύχει είναι η υποστήριξη της δημοκρατίας και η υποστήριξη των λαών της Τινησίας και της Αιγύπτου. Ευχαριστώ. Έξι προτάσεις ψηφίσματος για να κλείσει η συζήτηση, τελειώνει η συζήτηση και η ψηφοφορία θα γίνει αύριο στις 11.30.